Τελευταία στιγμή ε, έγινε αυτή η αλλαγή. Η κυρία Ματζόνη δεν θα μπορέσει να προεδρεύσει ε, στο πρώτο μέρος της συνεδρίασης, γι' αυτό και θα την αντικαταστήσω. Μόλις ε, διάβασα για ενημέρωσή μου το πρόγραμμα και τη μέση διάταξη, συγχωρήστε με αν κάνω κάποιο λάθος. Τώρα, η κυρία Αντζελίλη δεν θα έρθει στη συνεδρίασή μας. Έτσι και το σημείο 15 στην ημερήσια διάταξή σας μπορείτε να το διαγράψετε. Οπότε, το πρώτο θέμα είναι η ψηφοφορία. Ναι, ορίστε, ποιος θέλει το λόγο. κυρία ε, ε ναι, θέλω να σας πω κυρία Πρόεδρε ότι υπάρχει κάποια ανομαλία στα πρακτικά. Στα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης και ε, θα ήθελα να προτείνω κάποιες τροποποίησεις γραπτώς. Στα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης έχω ένα πρόβλημα. Θέλετε να το συζητήσουμε σήμερα. Όχι, όχι. Γραπτός, γραπτός θα υποβάλω κάποιες ε, τροποποίησεις. Ε, όταν θα φτάσουμε σε αυτό το θέμα θα το πείτε στην έγκριση των πρακτικών. Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη λοιπόν θα πρέπει να ξαναψηφίσουμε την έκθεση ε, για την ειδική έκθεση του κυρίου Διαμαντούρου ε, λόγω ενός τεχνικού προβλήματος κυρία τα διάφορα θα τα πούμε τώρα ή στο τέλος. Γιατί είχα μια πρόταση για τα διάφορα, γιατί θέλω μετάφραση για κάτι. Α, σε λίγα λεπτά. Να δούμε πρώτα ε, ποιο είναι το πρόγραμμά μας και μετά θα το συζητήσουμε. Θέλω να σας εξηγήσω για την ημερήσια διάταξη ότι λόγω ενός τεχνικού προβλήματος την τελευταία φορά που ψηφίσαμε για αυτή την ειδική έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητού είχαμε την παλιά εκδοχή. Γι' αυτό ήταν λάθος. Ε, και θεωρήσαμε ότι καλύτερο και απαραίτητο ήταν να ξαναψηφιστεί η νέα εκδοχή της έκθεσης σε περίπτωση που ε, κάτι ε, ήταν λάθος. Ελπίζω να διαβάσετε και τη σωστή, την πιο πρόσφατη και να θέλετε να ψηφίσετε εκτός αν δεν θέλετε να ψηφίσετε, να ξαναψηφίσετε. Δεν υπάρχουν τροπολογίες όμως και ε, για λόγους τυπικούς, ε, για να είμαστε τυπικώς εντάξει με την έκθεση αυτή που είναι πάρα πάρα πάρα πολύ σημαντική πρέπει να ξαναψηφίσουμε. Να συνεχίσουμε. Η βασική ε, ε, ιδέα της σημερινής συνεδρίασης αφορά ορισμένες ε, αναφορές για τα δικαιώματα των παιδιών και για την γονική μέρημνα και τη γονική ευθύνη. Ζητήθηκε την προηγούμενη φορά συζήτηση και έκθεση από τον καθηγητή Τζαμπάλο Ρωμάνο ο οποίος ε, παρευρίσκεται και θα μας παρουσιάσει την έκθεσή του. Καλώς ορίσατε. Ε, χαίρομαι που σας βλέπω εδώ και θα ε, αρχίσουμε από αυτό. Άλλη ενότητα αναφορών έχει να κάνει με τα ίδια προβλήματα, τα δικαιώματα των παιδιών και έχουμε και τους αναφερομένους ή εκπροσώπους τους παρόντες 8, 9 και 14 είναι θέματα τα οποία θα μας παρουσιαστούν κατόπιν επιλογής. Αργότερα, κατά τη διάρκεια του απογευματός, γύρω στις 6 παρατέταρτο, η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, κυρία Βίβιαν Ρέντινγκ, έχει προγραμματιστεί να έρθει για να μιλήσει για αυτό το θέμα, τα ειδικά ζητήματα των ε, παιδιών. Αύριο τώρα. Μετά τη συνεδρίαση των συντονιστών θα υπάρξει και περαιτέρω ευκαιρία να συζητήσουμε την ε, γνωμοδότηση Χάνκης για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όχι μόνο. Επίσης θα ακούσουμε και τον κύριο Βίλαντ για την πρόσφατη επιτροπή ε, που μετέβη στην Αυστρία. Γύρω στις 12 παρατέταρτο δηλαδή θα συζητηθούν τα αυριανά αυτά θέματα. Τον αναφορών δηλαδή θα μας παρουσιαστεί αναφορά 22 και επίσης και κάποιες άλλες που έχουν σχέση με το Βέλγιο 23 και 24. Έχετε σχόλια για την ημερησία διάταξη, παρακαλώ, ερωτήσεις. Ανακεφαλαιώνω. Η κυρία Αντζελίλη δεν θα έρθει, η κυρία Βιβιάν Ρέντινγκ θα έρθει στις 6 παρατέταρτο και αυτά είναι τα βασικά σημεία στην ημερησία διάταξη. Ας επανέλθουμε σε αυτό που είπε η κυρία Γκρινή προηγουμένως. Uh, για ε, την έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων της 29ης και 30 Σεπτεμβρίου. Η κυρία Γκρουνή, θα ήθελα απλώς να μην ψηφιστούν ως έχουν, να μην εγκριθούν τα πρακτικά ως έχουν, διότι θα ήθελα να γίνουν κάποιες τροποποίησεις τα πρακτικά που μας έχουν διανεμηθεί δεν ε, αντιστοιχούν στα όσα συζητήσαμε, ιδιαίτερα στις συνεδρίες των συντονιστών. Θα σας υποβάλω όμως γραπτός αυτές τις τροπολογίες μου. Χωρίς μικρόφωνο, κύριε Παλιαδέλη. Στην περίπτωση αυτή είναι καλύτερο να δούμε τις γραπτές σας ε, τροπολογίες που προτείνετε τροποποίηση των αρχικών ε, πρακτικών ή του κειμένου που σας έχει διανεμηθεί για να μην υπάρξει καμία παρεξήγηση. Η κυρία Άουκεν ήθελε να πει κάτι. Ναι, στα διάφορα σας είπα ότι ήθελα να θέσω κάτι. Ξέρω ότι είναι νωρί, αλλά μήπως θα το διεκπαιρώσουμε τώρα να τελειώνουμε. Ένα δελτίο τύπου ή και blog της κυρίας Μαζόνη του Σαββάτου αναφέρεται στην κατάσταση στην Καμπανία και είναι μόνο στα Ιταλικά. Και θα παρακαλούσα πάρα πολύ τα έγγραφα αυτά να τα λάβουμε και στα Αγγλικά πριν συνεδριάσουν αύριο οι συντονιστές. Δεν ξέρω αν είναι εφικτό κάτι τέτοιο, λέει η Πρόεδρος, ρωτώ με. Γιατί εξ όσων γνωρίζω, λέει η κυρία Άουκεν, είναι κρίσιμη σημασία σε σχέση με τα όσα έχουν συμβεί. Ένα προσχέδιο, κάτι, να δούμε, να καταλάβουμε τι λέει όμως, γιατί ε, συγκλονίστηκα όταν το διάβασα. Τώρα τι το διάβασα, έριξα μια ματιά, αλλά είναι φτωχά τα Ιταλικά μου. Και θα ήθελα πάρα πολύ να μεταφραστεί. Δηλαδή απόψε, πριν συνεδριάσουν αύριο το πρωί συντονιστέ. Ναι, θα παρακαλούσα πάρα πολύ αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Υπάρχει. Θα το ερευνήσουμε και θα σας πούμε. Δεν ξέρω, λέει η γραμματεία. Ε, εντάξει για να δούμε απλώς τι λέει αυτό το δελτίο τύπου και το blog. Έτσι ένα σχέδιο, μια σύνοψη, μια περίληψη, θέλετε. Not, not, not, not an accurate translation. Would you be satisfied with the points or something? Okay then. You know, I can see it's about our... Λοιπόν, είναι για την έκθεσή μας και έχω την αίσθηση ότι είναι και κατά της αντιπροσωπείας και ο πρόεδρος της ε, ε, αντιπροσωπείας που πήγαμε στην καμπανία, γιατί είναι και πρόεδρος, δεν είναι ένα τυχαίο μέλος της Επιτροπής μας. Ναι, ναι, κατανοώ απολύτως αυτό που λέτε, λέει η πρόεδρος. Γίνεται αυτή, ε, ε, ε, υπάρχει δυνατότητα έστω και μια μικρή περίληψη των βασικών σημείων. Καλώς. Τίποτα άλλο λοιπόν, uh, uh, συμφωνήθηκε. Λοιπόν, η 900 του 2007 και η 1792 του 2009, αυτές οι δύο θα ξανανοίξουν, έτσι έχει συμφωνηθεί νομίζω. Αντιθέτως, η 1768 του 2009 ενδεχομένως μπορεί να κλείσει. Εντάξει. Εάν δεν έχουμε τίποτα άλλο σχετικά με αυτά που σας ανακοινώνω, μπορούμε να περάσουμε στην ουσία των εργασιών. Δηλαδή στην ψήφιση της νέας εκδοχής της έκθεσης, της σωστής δηλαδή, της ορθής, της διορθωμένης, ε, για την ειδική έκθεση του κυρίου Διαμαντούρου. Θέλετε να ψηφίσουμε. Uh, not, not, ε. uh... So, raise your hands, those who agree. Η ψήφη υπέρ, παρακαλώ. And those who disagree. Κατά. Nobody. Nobody. Ουδής. Ομόφωνα μάλλον. Ε, καμιά αποχή, κάποιος που να διαφορεί. Όχι. Ευχαριστώ και πάλι όλους σας και για την προηγούμενη φορά και για τώρα. Λοιπόν, έχουμε τον καθηγητή τώρα που θα μας παρουσιάσει τη μελέτη για τη γονική μέρη. Ο καθηγητής κύριος Ρωμάνο, παρακαλώ. So, Professor Romano, are you ready to start with your... Είστε έτοιμοι, είστε έτοιμος κύριε καθηγητά. Θα μιλήσω γαλλικά, αν δεν σας πειράζει. Ε, Χωρίς μικρόφωνο ο κύριος Ρωμάνο. Α, το το μικρόφωνο. Ωραία, δουλεύει λοιπόν τώρα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Είμαστε εδώ για να σας παρουσιάσουμε τα πιο καυτά αποτελέσματα μίας μελέτης σχετικά με τη γονική ευθύνη και την κυδαιμονία των παιδιών ε, όταν έχουμε διασυνοριακά διαζύγια. Πριν από 1,5 χρόνο εμείς τελειώσαμε τη δουλειά μας, οπότε θα το έχετε δει είτε στα γαλλικά είτε στα αγγλικά. 250, 250 ε, σελίδες με δύο παραρτήματα. Πολύ σύντομα πώς διαρθρώνεται η μελέτη. Εμείς ε, Μαζέψαμε πρώτα απ' όλα τις στατιστικές βάσει της ισχύουσας μεθοδολογίας για το θέμα δηλαδή των διασυνοριακών διαζυγίων ανά την Ευρώπη. Δεύτερον, ε, κοιτάξαμε την ε, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία η οποία είναι άφθονη για να λάβουμε υπόψη μας αυτό, αυτή τη διάσταση των διασυνοριακών διαζυγίων. Και μετά ανάλυση και εθνικές νομοθεσίες. Ποιες είναι οι εθνικές πρακτικές. Σχετικά δηλαδή με το ποιος κρατάει τα παιδιά, ποιος έχει τη γονική μέρημνα και πώς οργανώνονται οι επισκέψεις. Και το τελευταίο τμήμα είναι ένας απολογισμός της πρόοδου που επιτεύχθηκε τα τελευταία χρόνια και αυτό λόγω μια σημαντικής παρέμβασης του, του Ευρωπαίου νομοθέτη, πρόκειται για το νόμο ε, Βρυξέλλες 2α, έτσι τον ονομάζουμε αυτόν τον νόμο στην ε, νομική αργό. Ποιες χώρες λάβαμε υπόψη μας ως δείγμα, δεν είχαμε και μεγάλες επιλογές δηλαδή, έπρεπε να Ξετάσουμε υποχρεωτικά την ε, Γερμανία και την ε, Γαλλία, την Ισπανία λόγω μεγέθους και όπως δείχνουν και οι στατιστικές ε, πρόκειται για μια χώρα όπου μεταφέρονται τα παιδιά, όχι πάντοτε νόμιμα. Πήραμε και την Πολωνία γιατί χρειαζόταν μια χώρα της Ανατολικής Ευρώπης λόγω μεγέθους. Το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν υποχρεωτικό ε, και τη Σουηδία τη διαλέξαμε, είχαμε δηλαδή επιλογή μεταξύ δύο σκανδιναβικών χωρών. Την Σουηδία την πήραμε και εδώ πάλι λόγω πληθυσμού. Μερικές τώρα έννοιες κλειδί πριν περάσουμε στις, στις ε, στατιστικές. Τι εστί ένας χωρισμός. Το, την σεπαρασιόν την ακούμε πάρα πολλές φορές, γιατί θεωρούμε είτε ως ακύρωση του γάμου ή πολλές ε, φορές χωρισμός σημαίνει χωρισμός του κοινού βίου. Όταν έχουμε δηλαδή ένα χωρισμό ζευγαριού, το οποίο δεν είναι παντρεμένο. Ζητήθηκε και ένας ορισμός ε, του, ε, του όρου διασυνοριακή διάσταση. και τον ε, ορισμό και εμείς τον ψάξαμε μέσα από τον κανονισμό Βρυξέλλες 2α. Θεωρείται λοιπόν ε, διασυνοριακή μία διάσταση όταν ε, ο αυτός ο οποίος έχει την γονική μέρημνα ή ισχυρίζεται ότι την έχει βρίσκεται μεταξύ δύο χωρών, το παιδί το ίδιο. Έχουμε είτε ενδοκινοτικές διαστάσεις, είτε διαστάσεις οι οποίες έχουν σχέση με δύο ή περισσότερα κράτη, με ένα ή περισσότερα συγγνώμη, ευρωπαϊκά κράτη και ένα εξωευρωπαϊκό κράτος. Αυτά. Λοιπόν, για να λάβουμε υπόψη μας αυτήν τη δεύτερη κατηγορία διαστάσεων που σίγουρα έχει έναν δεσμό με μία τρίτη χώρα, ας πούμε οι Ηνωμένε Πολιτείε ή η αργεντινη Α, για τη μετάφραση μιλάω πολύ γρήγορα. Και αφού είναι Ιταλός, ομιλητή, ε, Ιταλός είμαι και μου λένε ότι μιλάω γρήγορα. Η, Ιταλίδα βουλευτής, η Γαλλίδα βουλευτής του λέει ότι έχει δυσκολία να τον καταλάβει και στα γαλλικά. Λοιπόν, ναι, δικαιολογημένη λοιπόν η παρατήρησή σας. Λέει ο μιλητής συνεχίζοντας εξίσου γρήγορα. Λοιπόν, ποια είναι η γονική ευθύνη λοιπόν. Βασιστήκαμε λοιπόν στον ορισμό του κανονισμού 2α, ο οποίος δεν αναιρεί τις εθνικές νομοθεσίες, λέει τα ίδια πράγματα. Δηλαδή ηθικών πρόσωπων το οποίο αναλαμβάνει την κυδαιμονία του παιδιού, είτε ή γονείς, ένας από τους γονείς. Ένας δικαστής επίσης μπορεί η δικαστική δηλαδή απόφαση ή διοικητική απόφαση για την ανάθεση της γονικής ε, μέριμνας χωρίς την μεσολάβηση του δικαστή. Ας πούμε στην Ιρλανδία είχαμε μία απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Στην Ιρλανδία προβλέπεται, αν έχουμε ένα ζευγάρι μη παντρεμένο, ο πατέρας δεν έχει κανένα γονικό δικαίωμα. Δεν πρόκειται λοιπόν για νομοθετική ρύθμιση, αλλά για, πρόκειται για ένα αφηρημένο μέτρο. Και αυτή η υποχρέωση αφορά και το παιδί και τα αγαθά του παιδιού. Πιο συγκεκριμένα, Ποιο είναι το δικαίωμα κυδαιμονίας. Και αυτό βασίζεται στον ορισμό που έχουμε στο Βρυξέλλες 2α για την επιμέλεια. Δηλαδή όταν έχουμε διασυνοριακή διάσταση ε, αποφασίζεται ποιος έχει το δικαίωμα της επιμέλειας. Τώρα για το δικαίωμα επίσκεψης και εδώ έχουμε πάλι έναν ορισμό που τον παίρνουμε πάλι από το Διεθνές Δίκαιο. Είναι το δικαίωμα του να μπορεί κανείς να διατηρεί επαφή και προσωπικές σχέσεις με το παιδί. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό όταν έχουμε διασυνοριακή διάσταση. Δηλαδή να μπορεί κανείς να πηγαίνει το παιδί σε έναν άλλο τόπο εκτός του τόπου κατοικίας για να επισκεφθεί τον, γονέα, τον γονιό του που κατοικεί αλλού. Να δώσω το λόγο στη συνάδελφο για να σας πει τι γίνεται από στατιστικής πλευράς και, από και στα πλαίσια της εθνικής νομοθεσίας. Ευχαριστώ. Είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα να παίρνω το λόγο σήμερα. Συνεχίζω λοιπόν την αφήγηση και σας παρουσιάζω τα δύο πιο σημαντικά τμήματα της μελέτης, συλλογή και ανάλυση των στατιστικών και το τμήμα της μελέτης που αφορά στη νομική ανάλυση των εθνικών διατάξεων. Για την συλλογή των στατιστικών στοιχείων η επιλογή της ε, μεθόδου συλλογής ε, ορίζεται από το βασικό στόχο της μελέτης, δηλαδή να μελετήσουμε τις ιδιαιτερότητες της χορήγησης της επιμέλειας σε περίπτωση διασυνοριακών διαστάσεων και διαζυγίων. Εμείς μπορέσαμε λοιπόν να δούμε ψάχνοντας τα στοιχεία κατά πόσο τα κράτη-μέλη έχουν αυτά τα στοιχεία και έχουμε δύο τύπων πληροφόρηση. Τα στοιχεία γενικού χαρακτήρα, ε, και τα ειδικά στοιχεία για τον διασυνοριακό χαρακτήρα. Έχουμε την δικαστική, ε, τα δικαστικά στοιχεία και τα στοιχεία για τα διασύγια και επίσης το πώς λύνονται τα θέματα επιμέλειας σε περίπτωση διαζυγίου. Τώρα, για τις διοσυνοριακές διαστάσεις και χωρισμούς. Όταν οι δύο γονείς είτε κατοικούν σε διαφορετικές χώρες ή έχουν διαφορετική υπηκότητα. Θελήσαμε λοιπόν να δούμε τον αριθμό των διαζυγίων στο κάθε κράτος μέλος και να δώσουμε μία ποσοτική εκτίμηση των διασυνοριακών διαζυγίων. Μετά ψάξαμε να δούμε τις υποθέσεις εκείνες όπου λύθηκε το θέμα της επιμέλειας των παιδιών. Αυτό μας επέτρεψε λοιπόν να διαπιστώσουμε εάν το θέμα της επιμέλειας λύνεται με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με την περίπτωση. Αν είναι εσωτερική η περίπτωση ή διασυνοριακή περίπτωση. Χαρακτηριστικά λοιπόν των στοιχείων που αναλύσαμε σε ορισμένα κράτη όπως στη Γαλλία και στην Αγγλία οι στατιστικές για τις διασυνοριακές διαστάσεις δεν τα έχουμε. Σε αυτές τις χώρες το διασυνοριακό στοιχείο δεν διαφαίνεται στις στατιστικές είτε γιατί δεν το κατέγραψε κανείς είτε γιατί η υπηκότητα ή ο τόπος κατοικίας ενός από τους ενδιαφερόμενους δεν αναφέρεται. Δύσκολα λοιπόν μπορεί κανείς να το βρει αυτό στις δικαστικές αποφάσεις. Επίσης δύσκολα μπορεί να βρει κανείς ε, και με μετά τη διαδικασία του διαζυγίου ή της ε, διάστασης δεν έχουμε ίχνη για την κατοικία του παιδιού εκτός πια και αν υπάρχει απαγωγή. Όταν έχουμε στοιχεία, αυτά τα στοιχεία είναι ανεπαρκή. Δεν είναι ενιαία τα στοιχεία, δεν κάνουν διαχωρισμό μεταξύ της ευρωπαϊκής και μη ευρωπαϊκής ηθαγένειας των πρωταγωνιστών και διαφαίνεται περισσότερο η υπηκότητα του καθενός και όχι ο τόπος κατοικίας. Αυτό συμβαίνει στη Γερμανία, στη Γαλλία και στην Ισπανία. Και αυτό λοιπόν δεν μας επιτρέπει να εκτιμήσουμε τα αποτελέσματα αυτών των χωρισμών ως προς τον τόπο κατοικίας μετά από τη δίκη. Για το θέμα τώρα της επιμέλειας, τα στοιχεία πολλές φορές λείπουν. Αυτό λοιπόν μας εμποδίζει να εκτιμήσουμε το ρόλο του διασυνοριακού παράγοντα στο, ως προς την κατοικία των παιδιών. Μεταξύ των τάσεων εμείς ε, διαπιστώσαμε ότι έχουμε πολλούς μικτούς γάμους, ας πούμε στην Ισπανία και στη Γερμανία. Και στην Σουηδία πάνω από 20% των παιδιών έχουν ζήσει, έχουν βιώσει ένα διαζύγιο. Έχουμε επίσης αύξηση των διασυνοριακών διαζυγίων στην Πολωνία από τότε που η Πολωνία έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θέμα της κοινή επιμέλειας δεν το παρεμποδίζει η απόσταση ως προς την κατοικία των γονέων. Θέλαμε λοιπόν εμείς να δούμε αν η διασυνοριακή φύση της όλης υπόθεσης είχε επίδραση στην επίλυση της επιμέλειας των παιδιών. Και εδώ είναι σαφές το πράγμα. Ο διεθνής ή όχι χαρακτήρας της διαμάχης δεν φαίνεται να επιδρά στην δικαστική πρακτική για το θέμα. Τα στοιχεία που έχουμε δεν επικυρώνουν τη θέση ότι η υπηκότητα του γονιού επιδρά στην άσκηση της επιμέλειας ή των γονικών του, της γονικής μέρημνας. Δεν πρόκειται λοιπόν για αποφασιστικούς παράγοντες κρίσης. Τα στοιχεία επίσης που έχουμε δεν δείχνουν καμία τάση των εθνικών δικαστηρίων να βοηθούν τους δικούς τους υπηκόους για την επιμέλεια. Επίσης, λαμβάνεται υπόψη και η επιθυμία του παιδιού. Η στατιστική μελέτη που σας παρουσίασα συνοδεύεται από μια νομική και νομοθετική μελέτη σχετικά με τη γονική μέρημνα, την επιμέλεια, το δικαίωμα επίσκεψη σε περίπτωση διασυνοριακών διαζυγίων. Διαπίστωσε λοιπόν η μελέτη ότι η γονική μέρημνα η επι... ορίζεται αυτόματα από τη στιγμή που γεννιέται και αναγνωρίζεται το παιδί. Έχει γενικό χαρακτήρα, καλύπτει το παιδί και τα περιουσιακά του συμφέροντα. Τα, οι γονείς δεν μπορούν να αρνηθούν το δικαίωμα άσκησης της γονικής μέρημνας ούτε να την αναθέσουν σε τρίτο. Η γονική λοιπόν μέρημνα είναι ανεξάρτητη από τους δεσμούς των γονέων, είναι παντρεμένοι ή όχι. Μπορεί όμως αυτό το στοιχείο να παίξει ρόλο στην επιμέλεια. διαπιστώσαμε ότι οι γονικές συμφωνίες σε περίπτωση διάστασης εκτός από την Πολωνία είναι ενιαία με ορισμένες μικροδιαφορές όσον αφορά στην έννοια της γονικής μέρημνας στην Πολωνία, στη Γαλλία και στην Ισπανία τη γονική μέρημνα σε περίπτωση χωρισμού μπορούμε να τη δώσουμε αποκλειστικά, να την αναθέσουμε αποκλειστικά σε ένα γονιό. Στη Γερμανία όμως το παιδί μπορεί να φέρει αντίρρηση σε συμφωνία των γονιών και τότε ο δικαστής αποφασίζει για το πώς θα ασκηθεί αυτό το δικαίωμα. Για την επιμέλεια είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα της επιμέλειας. Γιατί η επιμέλεια ορίζεται μόνο όταν έχουμε διάσταση, ε, χωρισμό. Εκτός από τη Σουηδία, η ειδική έννοια της επιμέλειας υπάρχει σε όλα τα κράτη-μέλη. Ερμηνεύεται όμως διαφορετικά. Στην Γαλλία, στην Πολωνία και στο Ηνωμένο Βασίλειο η επιμέλεια ορίζει και την αρμοδιότητα του να αποφασίζει ο γονιός που, να μείνει, που θα μείνει το παιδί, χωρίς όμως να υποχρεώνει να κατοικεί μαζί με το παιδί. Στη Γερμανία η επιμέλεια λέει ότι πρέπει να ζει ο γονιός με το παιδί. Στην Σουηδία είναι εντελώς ανεξάρτητη από το θέμα του τόπου κατοικίας. Ως τώρα προς την ε, εναλλακτική επιμέλεια, όταν οι γονείς ε, κατοικούν διαφορετικά, μπορεί να έχει ο καθένας την ε, μέρημνα το, τμηματικά παντού εκτός από την Πολωνία για το δικαίωμα επίσκεψης δεν είναι μόνο δικαίωμα του γονιού που κατοικεί σε διαφορετικό τόπο από το παιδί, αλλά κυρίως είναι δικαίωμα του παιδιού για να, διατηρήσει το, να διατηρεί το δικαίωμα <coughs> σχέσεων με, τα, με τους δύο γονιούς σε περίπτωση διαζυγίου. Και είναι κοινή αυτή η αρχή σε όλα τα κράτη-μέλη που αναλύσαμε. Λίγες διαφορές έχουμε σε αυτή την έννοια. Η διαφορά βρίσκεται μόνο στο, καταναγκαστικό, καθαναγκασμό της επίσκεψης ή όχι. Είναι δικαίωμα ή δεν είναι δικαίωμα. Επίσης, ποιοι είναι οι δικαιούχοι του δικαίωματος επίσκεψης. Περιορίζεται στους γονιούς ή εφαρμόζεται επίσης σε άλλους, ας πούμε στους παππούδες. Τελευταίο σημείο η έννοια του συμφέροντος του παιδιού. Σε όλες τις αποφάσεις για τη μέρημνα, την επιμέλεια και την επίσκεψη σε περίπτωση χωρισμού των γονέων και ακόμη περισσότερο όταν έχουμε διασυνοριακή διάσταση. Βέβαια πρόκειται για μία έννοια αρκετά φλούος προς το πλαίσιο της που επιτρέπει να αναζητούμε τις πιο προσαρμοσμένες στις ανάγκες του παιδιού λύσεις ανάλογα με την περίπτωση. Ορισμένες νομοθεσίες όμως έχουν και ένα νομοθετικό ορισμό. Π.χ. στην Γαλλία το βασικό συμφέρον του παιδιού είναι να διασφαλίζεται η ευημερία του παιδιού. Στην Πολωνία λένε το προτζέσκα, ευημερία δηλαδή η ικανοποίηση των προσωπικών αναγκών και των περιουσιακών του αναγκών. Στην Σουηδία υπάρχει μία γενική διάταξη που ορίζεται συμφέρον των παιδιών και λέει και έχει να κάνει με την προστασία του παιδιού ε, κατά ιασδήποτε κατάχρησης ή κακομεταχείρισης και δεύτερο το παιδί να έχει σε περίπτωση χωρισμού μια στενή σχέση και με τους δυο γονιούς. Τώρα, οι νομολογίες, όλα τα κράτη που μελετήσαμε, δείχνει ότι καλύπτει και το δικαίωμα του παιδιού να εκφράζεται, κυρίως όταν οι γονείς έχουν διαφορές μεταξύ τους. Και αποτελεί μια κοινή αρχή σε όλα τα κράτη-μέλη. Τώρα το θέμα είναι ποια σημασία δίνεται στη βούληση του παιδιού και πώς ασκούνται τα δικαιώματα όπου έχουμε τις πολλές διαφορές σήμερα. Τα νομικά συστήματα τα οποία φαίνεται να δίνουν μεγάλη σημασία στο παιδί είναι η Γερμανία, η Σουηδία και, μερικά από και εδώ και μερικά χρόνια η Ισπανία. Δίνεται επίσης ιδιαίτερη σημασία στα συμφέροντα του παιδιού σε περίπτωση διασυνοριακής διάστασης. Για τα θέματα επιμέλειας, όταν αλλάζει κατοικία το παιδί και πάει στο εξωτερικό, αυτό δεν θεωρείται κατά του συμφέροντος του παιδιού, αυτή στιγμή πληρούνται ορισμένοι όροι. Η βασική έννοια η οποία ορίζει όλη αυτή την ε, διαδικασία είναι η αρχή της συνέχειας. Αυτό σημαίνει ότι η, κατοική, μετακόμιση του παιδιού στο εξωτερικό δεν σημαίνει ένα σπάσιμο με το κοινωνικό, τον κοινωνικό, αισθηματικό και γλωσσικό του περίγυρο. Επίσης, το δικαίωμα επίσκεψης του άλλου γονιού πρέπει να περιφρουρείται. Για το δικαίωμα τώρα επίσκεψης ή επισκέψεις του παιδιού του ιδίου προς το εξωτερικό δεν θεωρούνται κατά των συμφερόντων του παιδιού εκτός και αν υπάρχει εμφανής κίνδυνος απαγωγής στην Ισπανία ας πούμε ή αν η απόσταση είναι πολύ μεγάλη. Σουηδία. Αυτά σας ευχαριστώ. Και ξαναδίνω το λόγο στον καθηγητή κύριο Ρωμάνο. Επανερχόμεθα λοιπόν στο διεθνές επίπεδο μετά από αυτήν την ε, περιγραφή των στατιστικών και των εθνικών νομοθεσιών. Διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ εθνικών νομοθεσιών οι έννοιες διαφέρουν από τη μία χώρα στην άλλη, αλλά καταλήγουμε σε διαφορετικά αποτελέσματα όταν αυτές τις αρχές τις θέτουμε στην πράξη. Παίρνοντας εμείς λοιπόν όλα τα διεθνή κείμενα που ισχύουν σήμερα στην Ευρώπη, διαπιστώνουμε ποια είναι η διεθνής ρύθμιση και κυρίως η ευρωπαϊκή ρύθμιση που να είναι ικανοποιητική για όλα αυτά τα θέματα. Βέβαια, οι γονείς οι ίδιοι, το παιδί και όλοι όσοι ισχυρίζονται ότι έχουν δικαιώματα πάνω στο παιδί να μπορούν να προσφεύγουν στο δικαστήριο για να λαμβάνεται μια σαφής απόφαση εκτός και να έχουμε μια αλλαγή συγκυρίας για τα θέματα επιμέλειας και επίσκεψης. Θα πρέπει δε το περιεχόμενο και η εμβέλεια της απόφασης να είναι υπέρ του παιδιού, κυρίως, είναι το υπέρτατο συμφέρον, έτσι ορίζεται στα αγγλικά, Και εκεί πρέπει να λαμβάνεται η υπόψη κατά τη λήψη της απόφασης αυτό το συμφέρον του παιδιού σε περίπτωση δηλαδή διασυνοριακής διάστασης. Η άσκηση λοιπόν αυτών των δικαιωμάτων θα πρέπει να διαπιστώνεται επίσκεψη δηλαδή και επιμέλειας να διαπιστώνεται ότι ασκείται πραγματικά και να μην πλήττει τις κοινοτικέ ελευθερίες. Τώρα, ποιο είναι το κακό που πρέπει να καταπολεμήσουμε στην Ευρώπη και παγκοσμίω. Πρέπει να αποφύγουμε να έχουμε δύο διαφορετικές αποφάσεις πάνω στο ίδιο παιδί. Α, πάντα μου φέρνουν σημειώματα ότι μιλάω πολύ γρήγορα, δεν, έχω, δεν είμαι συνηθισμένος να την χάνω διερμηνίας, λέει ο μιλητής. Να, το 90 λοιπόν συνεχίζει ακάθεκτος, υπήρξε μία διμερής επιτροπή γερμανογαλλική όπου είχαμε μία γερμανική απόφαση και μία γαλλική απόφαση. Να, φανταστείτε εσείς ότι ο πατέρας είναι Γάλλος και η μαμά Γερμανίδα. Πρέπει να αποφύγουμε τα δύο δικαστήρια, ούτως ώστε να μην είναι το κάθε δικαστήριο χωριστά που θα αποφασίζει για τον καθένα. Διότι αν αποφασίσουν δύο δικαστήρια διαφορετικά μπορεί να έχουμε δύο διαφορετικές αποφάσεις. Π.χ. Ας πούμε οι Γάλλοι να αποφασίσουν ότι την επιμέλεια θα την έχει ο Γάλλος πατέρας. Και οι Γερμανοί να αποφασίσουν ότι την επιμέλεια θα την έχει η Γερμανίδα μητέρα. Και τότε έχουμε εδώ μία σύγκρουση αποφάσεων. Και τι γίνεται, είναι εντελώς παράλογο αυτό. Γιατί όταν έχουμε πολλές αποφάσεις το αποτέλεσμα είναι σαν να μην έχουμε καμία. Αφενός και οι γονείς αφετέρου τα παιδιά δεν έχουν ιδέα ποια είναι τα δικαιώματά τους. Απ' τη μια έχουμε την απόφαση που λέει, τη γαλλική που λέει ο πατέρας έχει το δικαίωμα επιμέλεια και απ' την άλλη έχουμε την ε, γερμανική απόφαση που λέει όχι είναι η μητέρα που πρέπει να τα ασκήσει. Λοιπόν το παιδί τι γίνεται όταν πρέπει κανείς να αποφασίσει δηλαδή σε ποιο σχολείο θα πάει το παιδί ή αν το παιδί πρέπει να χειρουργηθεί. Και εδώ πάλι διαφορετικές γνώμες. Η μητέρα η οποία έχει το δικαίωμα της λήψης της απόφασης λόγω της λήψης του, απόφασης του γερμανικού δικαστηρίου λέει ότι πρέπει να πάει σχολείο στη Γερμανία. Και η γαλλική απόφαση δίνει την ίδια εξουσία στον Γάλλο μπαμπά. Λοιπόν, Μα πρόκειται για μια ευρωπαϊκή απάρνηση απόδοσης δικαιοσύνης. Δεν δίνεται απάντηση από τα νομοθετικά συστήματα. Έχουμε αντιφατικές απαντήσεις. Και δεν μπορούμε εξ να λύσουμε εμείς αυτή την αντίφαση. Πρόκειται για ένα χώρο μη δικαίου. Πρόκειται για κάτι το δραματικό. Δηλαδή πραγματικά είναι μια δραματική αντίφαση. Εμείς δημιουργούμε σήμερα με το άρθρο 67 τη ε, της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναν ευρωπαϊκό δικαστικό ε, ε, χώρο δικαιοσύνης και εσωτερικών. Και βλέπουμε το παιδί να παίζεται μπαλάκι από τη μία χώρα στην άλλη χωρίς ποτέ να ξέρει κανεί ποιος έχει δικαιώματα πάνω στο παιδί και τελικά ο καυγάς μεταξύ γονέων γίνεται σύγκρουση μεταξύ νομικών ε, τάξεων, με, νομικών συστημάτων. Και αν κανένας δεν έχει την, και την εξουσία να λύσει τελεσίδικα αυτή τη λύση. Πρόκειται λοιπόν, το λέω προβοκατόρικα, μου είπαν ότι μπορώ να το πω προβοκατόρικα και να το γράψω προβοκατόρικα, αλλά λύνεται τελικά με το νόμο της ζούγκλας. Δηλαδή ο πιο επιθετικός γονιός, αυτός ο οποίος τσιρίζει πιο, πιο δυνατά, είναι αυτός ο οποίος θα καταστήσει στεβαστή την απόφαση του δικού του δικαστηρίου και θα καταπατήσει την απόφαση του άλλου γονιού. Και είναι τότε αναποτελεσματικές, καθίστανται αναποτελεσματικές οι ευρωπαϊκές ελευθερίες διότι αν ο γονιός ο οποίος έχει την εξουσία στη Γαλλία πάει με το παιδί του στη Γερμανία τότε δεν έχει πια κανένα δικαίωμα διότι έχει μπει στη γερμανική επικράτεια όπου εκεί διέπεται από τη γερμανική απόφαση την οποία, η οποία έχει αποφασίσει ότι έχει το δικαίωμα επιμέλειας η μαμά. Πώς λοιπόν έρεται όλη αυτή η δραματική κατάσταση. Πρέπει η απόφαση που λαμβάνεται να λαμβάνεται υπέρ των συμφερόντων του παιδιού. Οπότε για να διασφαλιστούν τα συμφέροντα του παιδιού πρέπει να υπάρχει ένας ρόλος αρμοδιότητας. Θα πρέπει ας πούμε μια ή δυο χώρες να είναι αρμόδιες ανάλογα με το που το παιδί βρίσκεται να υπάρχει δυνατότητα διαλόγου μεταξύ των δικαστών των χωρών τους οποίους, τις οποίες αφορά αυτή η κατάσταση και να βρίσκουν μία λύση η οποία να είναι βιώσιμη. Πρέπει να αποφύγουμε οπωσδήποτε τις παράλληλες διαδικασίες, διότι μόλις είπα προηγουμένως, αν έχουμε μία σύγκρουση αποφάσεων. Μία διαδικασία στη Γαλλία, μία στη Γερμανία και οι δύο να προχωρήσουν και να καταλήξουν σε μία απόφαση, τότε έχουμε αυτή, τις διπλές αποφάσεις με όλα τα επώδυνα αποτελέσματα που σας ανέφερα. Πρέπει επίσης να μειώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τις πιθανο, την πιθανότητα αναγνώρισης αυτών των αποφάσεων στα άλλα κράτη-μέλη. Διότι τι γίνεται. Ένα αναπόφευκτο αποτέλεσμα, ας πούμε αν η γαλλική απόφαση δεν είναι αναγνωρισμένη στη Γερμανία ή στην Ισπανία, αυτό υποχρεώνει τη Γερμανία ή την Ισπανία να ξαναδικάσουν, να προχωρήσουν σε μία νέα δίκη όπου τα θέματα της γονικής επιμέλειας να λύνονται διαφορετικά από τη μια χώρα στην άλλη. Τι υπάρχει σήμερα για να έχουμε μία ιδανική κατάσταση και να αποφύγουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Έχουμε πολλά μέσα. Ορισμένοι λένε ότι ίσως υπάρχουν και πάρα πολλά. Και γιατί και αυτό είναι ζημιογόνο. Διότι αν έχουμε πολλές διεθνείς συμβάσεις, αφενός συγχέονται οι δικαστές, αλλά και αυτά τα μέτρα, αυτά, αυτές οι συμβάσεις μπορεί να οδηγήσουν επίσης σε αντιφατική λήψη αποφάσεων. Πρόκειται επίση για μέτρα, αυτή, της, η σύμβαση της Χάγης και του Λουξεμβούργου του 81 είναι αρκετά ξεπερασμένα. Το μέλλον λοιπόν διαρθρώνεται μέσα από τρία μέσα. Σύμβαση της Χάγης του 80, με στόχο δηλαδή την καταπολέμηση των διεθνών απαγωγών παιδιών, του 96 πάντα της Χάγης, που είναι μια πλήρη σύμβαση, που εγκρίθηκε το 1996 αλλά άρχισε να ισχύει το 2002 σε ορισμένα κράτη, η Ευρωπαϊκή Ένωση επέτρεψε ορισμένα κράτη να υπογράψουν αυτή τη σύμβαση ορισμένα κράτη την υπέγραψαν άλλα όχι. Ας πούμε στη Γαλλία 1η Φεβρουαρίου θα αρχίσει να ισχύει, το 1η Φεβρουαρίου 2011, στην Πολωνία ισχύει εδώ και δύο χρόνια και πάει λέγοντας. Αλλά επίσης ένα μέσο το οποίο υπάρχει και το οποίο λειτουργεί αρκετά καλά και μπορούμε ίσως να το βελτιώσουμε είναι ο κανονισμός Βρυξέλλες 2α. Τώρα για τα ξεπερασμένα μέσα που έχουμε, να σας αναφέρω τις, ε, ε τις ατέλειες τους. Δεν σας, θα σας αναφέρω λοιπόν τα ξεπερασμένα μέτρα. Θα σας μιλήσω λοιπόν για τη Χάγη που έχει ως σκοπό την καταπολέμηση των απαγωγών παιδίων μεταξύ κρατών μελών. Πρόκειται για μία διάταξη που ισχύει παγκοσμίω, μία σύμβαση συγγνώμη, που ισχύει παγκοσμίω, δεν εφαρμόζεται μόνο στην Ευρώπη, σε 71-72 κράτη-μέλη εφαρμόζεται. Είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι Έχουμε όμως περιπτώσεις οι οποίες ε, οδηγούν σε άρνηση του παιδιού να επανέλθει στη χώρα και αυτό για λόγους που έχουν να κάνουν με την ενσωμάτωση του παιδιού, τη βούληση του παιδιού και τα λοιπά. Να μην σας πω τα τεχνικά τερτύπια διότι είναι πάρα πολλά. Μπορούμε όμως να βελτιώσουμε αυτή τη διάταξη για την επιστροφή. Και αυτή τη βελτίωση τη φέρνει ο κανονισμός της, των Βρυξελών. Τώρα, ο άλλος, η άλλη σύμβαση της ε, Χάγης είναι ένα μέσο ε, στη διάθεσή μας αρκετά πλήρες, αλλά υπάρχουν ακόμη αρκετοί λόγοι άρνησης αναγνώρισης της απόφασης. Και δεν υπάρχουν μέσα για την εκτέλεση, για τον καταναγκασμό στην εκτέλεση της απόφασης. Έχουμε λοιπόν τον κανονισμό Βρυξέλλες 2α που μπορεί να μας βοηθήσει να τροποποιήσουμε αυτό το μέσο. Πιο συγκεκριμένα στον τίτλο 513 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές οι διατάξεις επιτρέπουν από μόνες τους και ενθαρρύνουν την κοινότητα να παρεμβαίνει όταν πρέπει να διαμορφώσει, ένα, να δημιουργήσει ένα χώρο ελευθερίας, δικαιοσύνης και ασφάλειας. Ποια είναι λοιπόν τα μέσα που δίνουν αυτά τα άρθρα. Ε, πρέπει να τα ανασύρουμε για τη δική μας περίπτωση. Εμείς δεν θα πρέπει απλώς να απλουστεύσουμε την αμοιβαία αναγνώριση της απόφασης. Πρέπει πρώτα να οδηγήσουμε στην αναγνώριση την ίδια των αποφάσεων και την ε, σε την αναγνώριση των αποφάσεων για τη γονική μέρημνα. Και αυτό αποφεύγοντας την αντίφαση μεταξύ νομοθεσιών. Τώρα, Ποιες πρόοδους έχουμε από το 2000 και μετά. Έστω και αν τροποποιήθηκε βέβαια στο μεταξύ, γι' αυτό ονομάζεται Βρυξέλλες 2α. Συμπεριλαμβάνει λοιπόν αυτή η μεταρρύθμιση το κεφάλαιο που μας ενδιαφέρει πιο πολύ που είναι η γονική ευθύνη και το θέμα της μέρημνας. Αυτός ήταν ο περιορισμός, βασικό, το βασικό Αυτό ήταν το βασικό πρόβλημα του 102α στο παρελθόν, το θέμα της γονικής μέρημνας. Σήμερα οι πανεπιστημιακοί θεωρούν ότι είναι ένα μέσο το οποίο επιφέρει σημαντικές βελτιώσεις όχι μόνο ε, ως προς την κατάσταση του παρελθόντος αλλά ορίζει σαφείς κανόνες διότι η, την κύρια αρμοδιότητα την έχει η χώρα όπου κατοικεί το παιδί διότι πρώτα υπήρξε ένα πρόβλημα αρμοδιοτήτων μεταξύ της χώρας προέλευσης και της χώρας κατοικίας και υπήρχε το θέμα δηλαδή της αντίφασης Έτσι λοιπόν σήμερα υπάρχει ευελιξία όπου έχουμε δηλαδή ως επιλογή τη χώρα κατοικίας και υπάρχει επίσης η δυνατότητα να έχουμε έναν μηχανισμό μεταφοράς του ντοσιέ είτε ανάθεσης αυτού του ντοσιέ από τον τόπο κατοικίας σε μία άλλη αρχή για τη λήψη της απόφασης. Όσον αφορά τώρα το θέμα της λήψης της απόφασης, βλέπετε πόσο είναι επικίνδυνο όταν η απόφαση δεν λαμβάνεται. Σήμερα δεν υπάρχει πια αυτή η δυνατότητα σε τόσο μεγάλο βαθμό όσο στο παρελθόν. Ενοπίσαμε την διαδικασία του εξέκουο. Όταν έχουμε εμείς το θέμα της εκτέλεσης μίας απόφασης, απλουστεύεται το κοινοτικό δίκαιο. Και δεν είναι δαπανηρή η διαδικασία, είναι και γρήγορη. Και το θέμα της προστασίας του δικαιώματος επίσκεψης. Αυτό το δικαίωμα δεν ήταν επαρκώς σεβαστό στο παρελθόν. Ο νέος κανονισμός παρεμβαίνει σημαντικά και προβλέπει ότι εκείνο το τμήμα της απόφασης που αφορά στο δικαίωμα επίσκεψης θα πρέπει να γράφεται επίσημα και είναι αμέσως εκτελέσιμη υπάρχει εκτελέσιμη και στο άλλο κράτος μέλος. Υπάρχει δηλαδή η υποχρέωση. Τώρα, για τις πρόοδους που πρέπει να υπογραμμίσουμε, για τα θέματα απαγωγής των παιδιών. Εμείς είπαμε ότι η σύμβαση του 1980 εφαρμόζεται ικανοποιητικά αλλά υπήρχε πρόβλημα για τις, αποφάσεις, για αποφάσεις μη επιστροφή του παιδιού και ο κανονισμός στοχεύει στην καταπολέμηση αυτής της πλευράς και περιορίζει τους όρους επιβολής της επιστροφής του παιδιού Επίσης επιβάλλει και έναν πιο γρήγορο ρυθμό εκτέλεσης απόφασης, έξι εβδομάδες. Διότι αν δεν γίνουν σεβαστές οι έξι εβδομάδες πρέπει να δοθεί μία αιτιολόγηση για ποιο λόγο δηλαδή δεν κρατήθηκε η προθεσμία. Επιστροφής ή μη επιστροφής. Δεν μπορούμε εμείς να εμποδίσουμε την επιστροφή του παιδιού αν αποδείξουμε ότι στη χώρα στην οποία πρέπει να επιστρέψει το παιδί έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και τη διασφάλιση των συμφερόντων του παιδιού. Τώρα σε περίπτωση απαγωγής κάποιος πει όχι δεν το επιστρέφουμε το παιδί η χώρα προέλευσης του παιδιού μπορεί να λάβει η απόφαση που επιβάλλει την επάνωδο του παιδιού. Και τότε έχουμε αντίφαση. Η απόφαση όμως που θα υπερισχύσει μεταξύ των δύο ε, δικαστηρίων είναι η απόφαση του δικαστηρίου της χώρας προέλευσης του παιδιού. Κάτι άλλο το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον σε αυτόν τον κανονισμό είναι το θέμα της συνεργασίας των αρχών. Έχουμε τις κεντρικές αρχές οι οποίες θέλουν να διευκολύνουν τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών ε, για, την, ε, ε, για το πώς ζει το παιδί, για το πώς προστατεύονται τα συμφέροντά του. Και οι αρχές μπορούν να ασκήσουν αυτό το μέσο εποπτείας, το οποίο δεν είναι δαπανηρό, αυτό δεν ίσχυε στο παρελθόν. Μπορούμε επίσης να έχουμε πιο εύκολα διαμεσολαβητικές συμφωνίες και μπορεί λοιπόν η Ευρώπη να εκμεταλλευτεί αυτό το δικαστικό δίκτυο το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την ενίσχυση του διαλόγου που αναφέραμε προηγουμένως δηλαδή <coughs> τους διαλόγους μεταξύ δικαστικών αρχών. Λοιπόν, πώς βλέπουμε το μέλλον. Μπορούμε να έχουμε μία μεταρρύθμιση στο μέλλον. Πρόκειται για μία διαδικασία ε, ιδιαίτερα ε, λεπτή και μακρόχρονη και αρκετά βεβαρημένη θα έλεγα για την τροποποίηση διότι σήμερα είναι ακόμη δυνατό μία απόφαση η οποία αναθέτει την επιμέλεια δεν είναι εκτελέσιμη σε ένα άλλο κράτος και δεν αναγνωρίζεται, δεν είναι υποχρεωμένη, δεν είναι εκτελεστέα. Σε δέκα χρόνια ελπίζω ότι θα καταλήξουμε να φτάσουμε εκεί. Αλλά το τελευταίο βήμα το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι η υποχρεωτική αναγνώριση της επιμέλειας του παιδιού. Επίσης πρέπει να βρούμε μηχανισμούς ούτε ούτως ώστε να μην υπάρχει σύγκρουση αποφάσεων. Σας ανέφερα το παράδειγμα μεταξύ γερμανικών και γαλλικών αρχών. Επίσης πρέπει να βοηθήσουμε τη διαβούλευση μεταξύ των ενδιαφερομένων δικαστηρίων όταν η απόφαση αφορά ας πούμε στη Γερμανία και στη Γαλλία η απόφαση μπορεί να λαμβάνεται επίσημα από τη Γαλλία αλλά να υπάρχει υποχρέωση διαβούλευσης με το, με γερμανικό δικαστήριο. Υπάρχει βέβαια ένα πρόβλημα που είναι το πρόβλημα του συντονισμού μεταξύ του κανονισμού των Βρυξελών και της σύμβασης του 1996. Είναι ένα πολύ τεχνικό ζήτημα, δεν έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε γι' αυτό σήμερα. Για τις συστάσεις οι οποίες δεν θα οδηγούσαν σε τροποποίηση στο κείμενο των Βρυξελών μπορούμε να εναρμονίσουμε το θέμα της ακρόασης του παιδιού. Υπάρχουν ακόμη σημαντικές διαφορές για την ακροματικότητα του παιδιού μεταξύ των χωρών μελών και αυτό μπορεί να οδηγήσει στη μία αναγνώριση της απόφασης. Το να ακούγεται το παιδί στο γερμανικό δικαστήριο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί να οδηγήσει λοιπόν στη στη, στη Γερμανία συγγνώμη, σε μία μία αναγνώριση γαλλικής απόφασης που δεν έχει τόσο σημαντικό ρόλο το παιδί. Άλλη πρωτοβουλία που μπορούμε να αναλάβουμε είναι να ενθαρρύνουμε στην κατάρτιση εξειδικευμένων δικαστών είναι πολύ σημαντικό οι εθνικοί δικαστές να έχουν αρμοδιότητες ε, και κατάρτιση για, τα, ε, για στο διεθνές οικογενειακό δίκαιο και αυτά τα ζητήματα διεθνών διαμαχών να τα αναλαμβάνουν αυτοί οι ειδικά κατερτισμένοι δικαστές για το διεθνές δίκαιο. Επίσης το θέμα των ε, οικογενειακών συμβούλων και διαμεσολαβητών. Αυτά, ε, ε, αυτά, αυτά τα δίκτυα υπόσχονται πολλά. Θα μπορούσαμε λοιπόν εμείς να βασιστούμε και σε αυτά τα δίκτυα. Έχουμε μία οδηγία του 2008 που θα πρέπει να μεταφερθεί στο Εθνικό Δίκαιο μέχρι το 2011 σχετικά με τη διαμεσολάβηση. Αυτά. Νομίζω ότι είπαμε πάρα πολλά. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας και περιμένουμε τα σχόλιά σας και τις απαντήσεις σας. Ευχαριστούμε για αυτή την πολύ σημαντική μελέτη, η οποία αναδεικνύει ε, ναι, μια σειρά από προβλήματα με τα οποία ως Ευρωκοινοβούλιο θα έπρεπε να ασχολούμαστε λίγο πιο δυναμικά. Ε, θα δώσω όμως το λόγο στον συνάδελφο, τον κύριο Γιάρ και θα σας πω τις απόψεις μου στη συνέχεια. Ευχαριστώ. Äh, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση της μελέτης. Μπορεί να είναι περίεργο, παράξενο σας φανεί, αλλά παρόλα αυτά που μας είπατε δεν διευκρινίστηκαν τα πράγματα, δεν αποσαφινίστηκαν. Μπορεί να είναι περίεργο αυτό όταν το λέω εγώ, αλλά ε, είναι περίπλοκη η κατάσταση και τα θέματα των παιδιών, το δικαίωμα ε, να πηγαίνουν να γραφούν σε κάποια σχολεία και ε, οι διενέξεις μεταξύ των γονέων. Γιατί ε, όταν δεν συμφωνούν οι γονείς είναι δύσκολα τα πράγματα και όταν είναι μεγάλη η αντιπαράθεσή τους. Το είδαμε και από αναφορές που έρχονται στην Επιτροπή μας. Έχω μερικές ερωτήσεις που με ενδιαφέρουν. Θα κάνω όμως μία ερώτηση. Στο πρόβλημα Τη επιμέλεια. Ποιο έχει το δικαίωμα στο εσωτερικό όμω τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Περιορίζουμε σε αυτό. Ε, γιατί κάποια τάξη πρέπει να βάλουμε. Πρώτον, αν κατάλαβα καλά. Βέβαια, καλύτερα είναι πάντα να λύνονται τα πράγματα με φιλικού διακανονισμού και ειρηνικά, αλλά πολλέ φορέ καταλήγουν στα δικαστήρια και αυτό είναι αναπόφευκτο. Και χρειάζεται απόφαση δικαστική. Λοιπόν, κάτι που δεν κατάλαβα. Ποιο αποφασίζει, ποιο είναι αρμόδιο για να αποφασίσει γιατί λέτε ότι αυτό δεν είναι σαφώ ρυθμισμένο ή μήπω είναι. Ποιο αποφασίζει για την επιμέλεια, έχει λυθεί αυτό ξεκάθαρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μονοσήμαντα ή όχι. Ποιο είναι το δικαστήριο που έχει τη δικαιοδοσία να αποφασίσει. Και έρχεται η δεύτερη ερώτηση που θέσατε κι εσείς. Έστω ότι έχει αποφασίσει ένα δικαστήριο. Οι υπόλοιπε χώρες, κράτη-μέλη, εν πάση περιπτώσει, τη ενωση ε, είναι υποχρεωμένα να αναγνωρίσουν τη δεσμευτικότητα αυτής της απόφασης νέου. Και τρίτη ερώτηση. Λέτε στη μελέτη σας ότι υπάρχει μεν νομική οδός και αποφασίζεται, αλλά καμιά φορά ε, αυτό είναι εις βάρος των δικαιωμάτων των παιδιών, γιατί διαφέρουν οι αποφάσεις από χώρα σε χώρα σε ορισμένες χώρες προέχει το δικαίωμα και το συμφέρον των παιδιών, αλλά δεν ισχύει παντού αυτό. Και τελευταία ερώτηση. Στα κράτη-μέλη πιστεύετε εσείς ότι η δικαιοδοσία, η νομική βάση διαφέρει τόσο πολύ από χώρα σε χώρα, έτσι ώστε να χρειάζεται εναρμόνιση ή να επιδιώκουμε εμείς την εναρμόνιση. Και αν ναι, σε ποιους τομείς θα πρέπει να γίνει αυτή η εναρμόνιση. Αυτά. Ζητώ συγγνώμη, εγώ νομικό δεν είμαι. Μπορεί με ορισμένες ερωτήσεις να ε, σας φαίνονται ε, αδρές, έτσι, χοντρές, όχι ιδιαίτερα λεπτομερεί, αλλά είναι ένα θέμα που στην Επιτροπή Αναφορών έρχεται συχνά και πολύ συναισθηματικά φορτισμένο. Και το δικαστήριο, ε, καμιά φορά παίρνουν αποφάσεις στα δικαστήρια δικαστικές, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι απονέμουν δίκαιο ότι δικαιώνεται ο κόσμος δηλαδή επειδή ε, εφαρμόζεται κάποιο νόμο. Και στο μέλλον θα μας αποσχολήσει πολύ περισσότερο αυτό. Ευχαριστώ. Ρωμάνο, θα σα παρακαλούσα να είστε σύντομο στην απάντηση σε αυτόν τον τεράστιο αριθμό ερωτήσεων και μεγάλων ζητημάτων που έθεσε ο κύριος Γιάρ. Ε, αν μπορείτε, γιατί έχουμε ε, κι άλλοι. Euh, σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Ερωτήσεις οι οποίες είναι πολύ ακριβείς Θα ξεκινήσω με το ζήτημα της αρμοδιότητα, της δικαιοδοσία. Είπατε, μας ρωτήσατε αν υπάρχουν ξεκάθαροι κανόνες δικαιοδοσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η απάντηση είναι ναι. Υπάρχουν κανόνες οι οποίοι είναι αρκετά σαφεί αλλά και ευέλικτοι. Και αυτό γιατί θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να εγγυηθούμε ένα ελάχιστο ευελιξία, τουλάχιστον όσον αφορά του κανόνε δικαιοδοσία μέσω των οποίων θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε συγκεκριμένα μία υπόθεση. Υπάρχει ένας γενικός βασικός κανόνας όσον αφορά την γενική δικαιοδοσία του κράτους ε, συνήθους ε, εγκατάστασης διαμονής του παιδιού. Αυτός είναι ο βασικός κανόνας. Αν όμως οι δικαστικέ αρχές θεωρούν ότι είναι σκόπιμο, μπορεί να μεταφερθεί η δικαιοδοσία προ τι αρχέ εκείνε που μπορεί να βρίσκονται εκτό του κράτου προέλευση. Θα μπορούσε να είναι το κράτο τη υπηκότητα του παιδιού, το κράτο τη περιουσία του παιδιού και το καθεξής. Υπάρχει δηλαδή δυνατότητα μεταφορά τη δικαιοδοσία. Μεταφορά τη δικαιοδοσία προ μια άλλη πιο κατάλληλη αρχή. Υπάρχει πάντω ένα βασικό κανόνα, μια βασική δομή όσον αφορά τη δικαιοδοσία. Και είχαμε στο παρελθόν και κάποιε περιπτώσει μεταφορά ε, τη δικαιοδοσία, η οποία όμω θα πρέπει να γίνει αποδεκτή από την αρχή εκείνη που θα δεκτεί τη δικαιοδοσία. Σε αντίθετη περίπτωση, η δικαιοδοσία παραμένει στην χώρα συνήθους διαμονής του παιδιού. Και ανοίγω και μία παρένθεση αυτή τη στιγμή. Συνήθις διαμονή, τι σημαίνει αυτό. Θα πρέπει να εντοπιστεί ποια είναι η συνήθις διαμονή. δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο ορισμός ε, για την ε, διαμονή αυτή. Γίνεται πάντω αναφορά στι διεθνεί ε, συμβάσεις. Προσπαθούμε να μην ορίσουμε όμω συγκεκριμένα τη συνήθη διαμονή, εναπόκειται πολύ συχνά στα δικαστήρια, στους δικαστές να δώσουν έναν ορισμό. Ο ορισμό ο παρέχεται αυτή τη στιγμή από τι Εθνεί Συμβάσει είναι αρκετά γενικό προκειμένου να επιτρέπει στι Εθνικέ Δικαστικέ Αρχέ να ορίζουν κατά περίπτωση καλύτερα το ζήτημα τη συνήθου διαμονή. Τώρα, υποχρέωση αναγνώριση μια δικαστική απόφαση. Υπάρχει το θέμα αυτό και πώ διευθετείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Α πούμε ότι έχουμε μια δικαστική απόφαση. Αυτή η δικαστική απόφαση μπορεί να κυκλοφορήσει ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η ερώτησή σας. Η απάντησή σας πάλι δεν μπορεί να είναι ναι ή όχι. Δεν υπάρχει υποχρέωση αναγνώρισης. Δεν υπάρχει υποχρέωση αναγνώρισης. Και θα ήθελα να διευκρινίσω εδώ πέρα όσον αφορά το δικαίωμα επιμέλειας. Υπάρχει όμως υποχρέωση αναγνώρισης όσον αφορά το δικαίωμα επίσκεψης στην περίπτωση αυτή και το δικαίωμα επίσκεψη, έχει ληφθεί μια δικαστική απόφαση π.χ. από τη Γερμανία, τότε αυτή μπορεί να εφαρμοστεί και να εκτελεστεί οπουδήποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί δηλαδή καμία δικαστική αρχή άλλη, πέρα από τη γερμανική προφανώ που έχει προχωρήσει στην απόφαση, να αντιταχθεί σε αυτή τη δικαστική απόφαση. Για την επιμέλεια όμω των παιδιών δεν υπάρχει ακόμα αναγνώρι... Ε, υποχρέωση αναγνώριση δικαστική απόφαση. Και αυτό γιατί υπάρχουν ακόμα κάποιοι λόγοι, ένα κατάλογο λόγων, έξι-εφτά λόγοι, για του οποίου μπορούμε να αρνηθούμε την εφαρμογή μια τέτοια απόφαση. Ας πάρουμε πάλι το παράδειγμα της γερμανικής απόφασης που θα μπορούσε να τύχει άρνηση, για παράδειγμα, στην Γαλλία. Η Γαλλία θα μπορούσε να αρνηθεί να γνωρίσει την απόφαση αυτή γιατί ενδεχομένως να μην ε, έχουν ε, καταφέρει να συμμετέχουν στην ε, δίκη όλοι οι συμβαλόμενοι, όλοι έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν ή μπορεί να μην έχει ακουστεί το ίδιο το παιδί. Μπορούμε να έχουμε βέβαια μία δικαστική απόφαση στην Γαλλία στην οποία δεν έχει ακουστεί το παιδί. Η δικαστική αυτή απόφαση παραμένει βέβαια γαλλική και δεν υπάρχει υποχρέωση αναγνώρισή τη στη Γερμανία. Ή μπορεί να υπάρχει μια συνεννόηση μεταξύ των δύο δικαστικών αρχών Γερμανία και Γαλλία. Εκτό μικροφώνη, Πρόεδρος. Θα πρέπει να είστε πολύ πιο σύντομο στι απαντήσει σα και εσεί πιο σύντομο θα θέτετε ερωτήσει. Το πρόβλημα είναι πολύ σημαντικό και υπάρχουν και πολλοί άλλοι συνάδελφοι που θα ήθελα αυτή τη στιγμή να υποβάλουν ερωτήσει. Και πρέπει να ακούσουμε επίση και τι αναφορέ και νομίζω ότι και αυτέ θα μπορούσαν να συμβάλλουν στο να καταλάβουμε καλύτερα την μελέτη σα, κύριε Τζανπάολο Ρωμάνο. Δεν ξέρω λοιπόν, μπορείτε να μα δώσετε μια σύντομη απόφαση και προφανώ μπορείτε να μείνετε κατά τη διάρκεια όλη τη συνεδρίαση. Το τρίτο ερώτημά σας τώρα, λέει ο κύριος Ρωμάνο, έχει να κάνει με την διακριτική μεταχείριση. Αναλύοντας την ομολογία, δεν μπορούμε να πούμε ότι οι εθνικές δικαστικές αρχές προχωρούν σε διακριτική μεταχείριση με βάση την ηθαγένεια, την πικότητα του παιδιού, των γονιών ή το τόπο διαμονής. Δεν νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να μιλάμε για μια διακριτική μεταχείριση. De facto μπορεί να υπάρχει μια διακριτική μεταχείριση αν θέλετε, γιατί ε, το παιδί μπορεί να μένει σε μια συγκεκριμένη χώρα, σε ένα συγκεκριμένο τόπο, μπορεί να επιθυμεί το παιδί να παραμείνει στη χώρα αυτή, να παραμείνει στη χώρα που διαμένει ένας από τους δύο γονείς, για παράδειγμα. Η τέταρτη ερώτησή σα ήταν και πιο δύσκολη και πιο πολύπλοκη. Δυστυχώ δεν μπορώ να απαντήσω με πάρα πολλέ λεπτομέρειε. Μα ρωτήσατε αν θέλουμε να εναρμονίσουμε το ζήτημα της γονικής μέρημνας. Υπάρχουν διαφορές αυτή τη στιγμή σημαντικές από τη μία χώρα στην άλλη. Θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε μία εναρμόνιση, σε κάποιους τουλάχιστον τομείς. Εγώ πιστεύω και το έχω προτείνει άλλωστε να ξεκινήσουμε με μία ακρόαση του παιδιού, δηλαδή να δούμε τις περιπτώσεις εκείνες που θα είχαν να κάνουν με την αναγνώριση αποφάσεων στις, ε, διασυνοριακές αν θέλετε υποθέσεις. Να δούμε δηλαδή αν μπορεί το ζήτημα της ε, μαρτυρίας του παιδιού της ε, να εισακουστεί ουσιαστικά το παιδί και να ισχύει αυτό έπειτα σε αποφάσεις, να ισχύει διασυνοριακά σε δικαστικές αποφάσεις. Εκτός μικροφώνου, Πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε πολύ. <laughs> Ήθελα να σας ευχαριστώ και όλους που ολοκληρώσετε την απάντησή σας. Θέλετε να προσθέσετε όμως προφανώς κάτι, έτσι δεν είναι. Ναι, σας ευχαριστώ. Καταλαβαίνω τα γερμανικά. Έχω ένα μικρό πρόβλημα. Δεν μπορώ να ακούσω την διερμηνία. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί το σύστημα. Δεν μπορούσα να ακούσω αυτά τα οποία είπατε εσείς τα ελληνικά. Πρέπει να επιλέξετε τη γλώσσα που θέλετε να ακούσετε στο κουμπί που υπάρχει εκεί πέρα, το μικρό κουμπάκι. Ε, σχετικά με την εισήγηση του κυρίου Ρωμάνο είναι η κυρία που θα ήθελε λάβετε υπόψη σας ότι έχουμε petitions που τις περιμένουμε αμέσως μετά. Παρακαλώ να είστε σύντομοι συνάδελφοι. Καταρχά να πω το εξή εισαγωγικά. Ε, για να καταλάβουμε αυτή την περιπλοκότητα των διεθνών προβλημάτων και να μπορέσουμε να τα λύσουμε, θα ήταν ε, ίσω σωστό να σκεφτούμε μήπω σε κάθε χώρα να υπάρχει ένα συνήγορο του παιδιού συνήγορος που είναι ε, δικηγόροι ε, και ασχολούνται με παιδιά και ε, με εφήβους τελείως ανεξάρτητη αρχή που βοηθάει και τα παιδιά και μπορούν τα παιδιά από μόνα τους να προσφεύγουν στο συνήγορο του παιδιού και για να μπορέσουμε καν να λύσουμε και να καταλάβουμε αυτά τα προβλήματα. Αυτό ευχαριστώ πολύ. Are you ready to... Μπορείτε να απαντήσετε, είστε έτοιμος. Στα γερμανικά. Όχι, όχι, μια στιγμή. No, no, ε, δεν έχετε το λόγο αυτή τη στιγμή. Περιμένουμε μία απάνταση. Θα έρθει και η σειρά σα. Απαντήστε, παρακαλώ πολύ, στην ερώτηση της κυρίας Βέρτμαν. Μπορεί να την ξαναπεί την ερώτηση γιατί δεν μπόρεσε να την ακούσε. Έκλεινα το μικρόφωνο εκείνη τη στιγμή. Μπορεί της παρακαλώ πολύ να επαναλάβετε στον κύριο Ρωμάνο σύντομα την ερώτησή σας. Λοιπόν, στη δική μου πατρίδα υπάρχει μια αρχή που λέγεται συνήγορος του παιδιού και του εφήβου. Ε, με ουδετερότητα, με ανεξαρτησία και μπορούν τα παιδιά και οι ανήλικοι να απευθύνονται για να εισακούονται σε αυτή την αρχή. Και θα ήθελα παρακαλώ σε όλη την Ευρώπη να υπάρξει αυτή η αρχή, η ανεξάρτητη αρχή για να έχουν το λόγο και τα παιδιά, για να λυθούν και αυτά τα τόσο περίπλοκα ε, προβλήματα. Τι ισχύει πού. l'institution euh, Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Καταλαβαίνουμε πολύ καλά ποιο είναι το νόημα της ερώτησής αυτής. Δυστυχώς όμως η ερώτηση αυτή ε, είναι εκτός του πεδίου εφαρμογή της δικής μας μελέτης. Δεν ασχοληθήκαμε άμεσα με την ερώτηση αυτή. Όσον αφορά τις ε, εθνικές πρακτικές. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι σε εθνικό επίπεδο υπάρχουν τέτοιες πρωτοβουλίες. Για παράδειγμα στη Γαλλία υπήρχε τουλάχιστον στο παρελθόν μέχρι πέρυσι, αν δεν κάνω λάθος, ένας συνήγορος, εθνικός συνήγορος για το παιδί, ο οποίος όντως έδινε τη δυνατότητα στο παιδί να ακουστεί για λόγους θεσμικούς και οργανωτικούς ο θεσμός αυτός ετέθην κινδύνο, το οποίο πραγματικά είναι κρίμα. Δεν ξέρω βέβαια αν σε κοινοτικό επίπεδο θα μπορούσαμε να είχαμε γενικευμένη μία τέτοια αρχή, ένα τέτοιο θεσμό. Θα έλεγα πάντως σε σχέση με την ερώτησή σας ότι όντως ναι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η πρακτική αυτή είναι καλή και θετική και μια μελέτη σαν τη δικιά μας θα μπορούσε να αποτελέσει μια απογραφή των βέλτιστων πρακτικών. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να αναλύσουμε, αν θέλετε, κάπω πρακτικέ που υφίστανται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένω, κάποιε θετικέ πρωτοβουλίε θα μπορούσαν να αποτελέσουν ε, τμήμα ενό καταλόγου. Εμεί αυτή τη στιγμή αναφερόμαστε σε πρωτοβουλίε που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε εθνικό επίπεδο. Για ποιο λόγο να μην προχωρήσουμε περισσότερο στην εφαρμογή θετικών πρακτικών από άλλε χώρε. Για ποιο λόγο να μην προσπαθήσουμε να θεραπεύσουμε, αν θέλετε, κενά και προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση όντω να αποτελέσει το χώρο εκείνο που θα διοχετεύονται περισσότερο οι θετικέ εθνικέ πρακτικέ. Μια διευκρίνηση ότι δεν μπορούν να πάρουν το λόγο παρά μόνο οι εκπρόσωποι ή οι ίδιοι οι καταγγέλλοντες ε, σε ό,τι αφορά τη διαδικασία και να παραδώσω την Προεδρία στην κυρία Ματσόνη που έχει έρθει πριν από λίγο. Σας ευχαριστώ. Buonasera. Allora, eh... Καλησπέρα. Μου είπανε ότι είμαστε στην πρώτη αναφορά στο σημείο 7. Δεν είναι παρόν ο εισηγητής, άρα το λόγο θα πάρει ο Μάρκου Ζαλεύσκη το λόγο, εκπρόσωπος της Κομισιόν. Good afternoon, Madam Chair. Καλησπέρα σας, κυρία Πρόεδρε, μέλη της Επιτροπής Αναφορών. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω που προσκαλέσατε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην σημερινή σας συνεδρίαση. Εκπροσωπώ την μονάδα που έχει να κάνει με τη δικαστική συνεργασία ε, όσον αφορά τις αστικές υποθέσεις. Θα πρέπει να σας ζητήσω συγγνώμη εξ ονόματος του επικεφαλής της μονάδας μου. Σήμερα είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα Τη αστική δικαιοσύνη, επομένω, η επικεφαλή μου βρίσκεται στη Σλοβενία και θα αναφερθεί σε κάποια από τα ζητήματα που θα καλύψουμε και σήμερα το απόγευμα. Είδατε, φαντάζομαι, την γραπτή μα απάντηση, τι γραπτέ μα παρατηρήσει που τροποποιήθηκαν μία φορά γιατί υποβλήθησαν για κάποια επιπλέον έγγραφα. Όπω θα δείτε από τι παρατηρήσει μα υπάρχουν τρία στοιχεία στα οποία αναφέρονται οι αναφέροντε. Το ένα έχει να κάνει με το ποινικό δίκαιο, το δεύτερο αναφέρεται στην δικαστική συνεργασία, που είναι το βασικό μέσο, αν θέλετε, που το επιδιοθέτουμε, και τρίτον, γίνεται αναφορά στην νομική αρρωγή. Εξετάσαμε και τις τρεις πτυχές και θα δείτε από το συμπέρασμά μας ότι όλα τα θέματα τα οποία θίγονται από τους αναφέροντες δεν εμπίπτουν στο κοινοτικό δίκαιο ή ακόμα και όταν εμπίπτουν στο κοινοτικό δίκαιο και πάλι είναι οι εθνικές αρχές εκείνες οι οποίες θα πρέπει να εφαρμόσουν την εθνική νομοθεσία σε συγκεκριμένε περιπτώσεις και πιο συγκεκριμένα σε περιπτώσεις ε, εκείνες που έχουν να κάνουν με την ε, μη παροχή νομικής αρρωγής στις οποίες αναφέρονται οι ε, αναφέροντες. Δεν θα ήθελα εδώ πέρα να μακρηγορήσω περισσότερο. Είμαστε προφανώ στη διάθεσή σα για να απαντήσουμε σε συγκεκριμένε ερωτήσει για τι περιπτώσει αυτέ και για άλλη μια φορά σα ευχαριστούμε πολύ που μα προσκαλέσατε. Θέλει κανεί το λόγο. Όχι. Κλείνουμε λοιπόν αυτή την αναφορά κατόπιν της απαντήσεως της Κομισιόν. Σημείο 8 είναι η αναφορά της Μαρινέλα Κολούμπο. Και είναι παρόν εδώ ο δικηγόρος και έχει το λόγο. Ή δικηγόρος. Θα κοιτάξω να είμαι όσο το δυνατόν πιο σύντομη. Πρέπει να σας πω ότι η αναφορά η οποία ε, ε, έχει προσυπογραφεί από 2.000 και πάνω ε, υπογράφοντες και όχι 134. Έχουν σταλεί σχετικές υπογραφές. Λοιπόν, η αναφορά αναφέρεται στην προβληματική του Jugendamt που είναι γνωστή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το θέμα επανετέθη πρόσφατα από την θέση της Ευρωβουλευτού της κυρίας Ναταλή Γκρίσμπεκ, την οποία την ευχαριστώ πολύ. Είναι γνωστό ότι κάθε κράτος Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει την αυτονομία του σχετικά με το οικογενειακό δίκαιο. Όμως είναι επίσης σαφές ότι κάθε κράτος της Ένωσης θα πρέπει να σέβεται τις διεθνείς και κοινοτικές νομοθεσίες και τις ε, σύμβασεις, όπως είναι η Σύμβαση της Νέας Υόρκης για το δικαίωμα των ανηλίκων παιδιών. Όπως ε, επίσης και τον κανονισμό των Βρυξελών 2α ε, που αναγνωρίζεται ότι θα πρέπει να, σε, να γίνονται σεβαστό το, τα δικαιώματα του παιδιού, τα πολιτιστικά του δικαιώματα όπως ε, και των διαφορετικών πολιτιστικών καταγωγών του παιδιού. Αναφέρομαι λοιπόν και στον κανονισμό, είπαμε, ε, Βρυξέλλες 2α και στην Σύμβαση της Χάγης του 1980 και στο άρθρο 21 της Συνθήκης ε, για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εγγυάται την ελεύθερη κυκλοφορία των Ευρωπαίων πολιτών. Η κυρία Κολόμπο υπογραμμίζει τις παραβιάσεις τις οποίες θεωρεί ότι υπέστη από τις γερμανικές αρχές τις διατάξεις που προανέφερα. Και αυτό λόγω του Kindeswohl που έχει να κάνει όχι με το ενδιαφερόν του παιδιού όπως το εννοούμε στην, ε, γενικώ στην Ευρώπη αλλά στο να παραμείνει το παιδί στην ευρωπαϊκή επικράτεια. Επίσης αυτό το Kindeswohl ασκείται μέσω της οργάνωσης Jugendamt που δεν είναι κοινωνική υπηρεσία διότι υπάρχει στη Γερμανία η Social Amt. <coughs> λοιπόν να σας πούμε τι είναι Jugendamt. Πρόκειται για ένα εθνικό γραφείο επιτήρησης της ε, ε, ε, γονικής κατάστασης και μπορεί να παρουσιάζει και να καταθέτει μάλλον καταγγελίες πράγμα το οποίο δεν ισχύει αλλού και παρεμβαίνει αυτόματα άσχετα από τα θέματα γονικής έρευνας και το Jugendamt τα δρά πάντοτε υπέρ του Γερμανού υπήκοου. Στην περίπτωση της κυρίας Κολόμπο, να σας πω τα παραδείγματα. Απαγορεύθηκε στην κυρία Κολόμπο να μιλάει Ιταλικά με τα παιδιά της. Ο υπάλληλος του Jugendamt, ο κύριος Μπόσλερ, δήλωσε το εξής το να αναγνωρίζεται κανείς ως Γερμανός εξαιτίας ε, της προφοράς μπορεί να οδηγήσει στην απόρριψη του παιδιού από την κοινότητα, από τη σχολική κοινότητα στην Ιταλία στην προκειμένη περίπτωση. Ε, επίσης το θέμα της διατροφής ε, επέπεσε στην ευθύνη της ε, κυρίας Κολόμπο και όχι στους δύο γονείς. Το Jugendamt έχει, έχει λάβει έχει αποφασίσει μάλλον μόνο σε συνεργασία με τον Γερμανό γονέα και δεν μπόρεσε η κυρία Κολόμπο να έχει πρόσβαση στον ντοσιέ της και αυτό γιατί αναφέρθηκαν ε, αρχές ε, privacy. Επίσης πάντοτε μέσα από αυτήν την περίεργη θέση το Jugendamt προβλέπει προληπτικά στις 24 Αυγούστου έγινε αυτό όταν ήταν στη Γερμανία να γραφτεί στις, ε, στους καταλόγους της Interpol λέγοντας ότι η κυρία Κολόμπο θα μπορούσε να φύγει από τη χώρα με ή χωρίς τα παιδιά και διαβάζουμε στα πρακτικά της δίκης. Υπάρχει κίνδυνος στα παιδιά της κυρίας Κολόμπο να μην έχουν καμία επαφή με τον πατέρα τους αν αυτή μετακομίσει στην Ιταλία και ο πατέρας δεν θα μπορέσει να ασκεί το δικαίωμα επίσκεψης. Το υπογραμμίζουμε αυτό γιατί βρίσκεται και στην ε, σύμβαση της Χάγης την επόμενη της, ε, του επαναπατρισμού της κυρίας Κολόμπο δεν είχαν τα παιδιά το δικαίωμα να μιλήσουν καν στο τηλέφωνο με τη μητέρα τους για δέκα μήνες και βάσει του Κίντεσβολ θεωρήθηκε ότι δεν μπορούσαν να ακούσουν ούτε καν από το τηλέφωνο τη μαμά τους η οποία συνελήφθη με το ένταλμα το οποίο σας προανέφερα. Ρωτώ λοιπόν πρώτον τι εστί, Κίντεσβολ, Ευθυγραμμίζεται αυτό με την έννοια των συμφερόντων του παιδιού. Δεύτερον, να σημάνω τον κόδωνα του συναγερμού. Αν εμείς θέλουμε να μπερδεύουμε το δικαίωμα της επιμέλειας με το δικαίωμα επίσκεψης, τότε στρεβλώνουμε και το αντικείμενο του κανονισμού Βρυξελών 2α. Και στην σύμβαση της Χάγης του 80 ξέρουμε ότι ο επαναπατρισμός γίνεται καταναγκαστικά μόνο όταν παραβιάζονται δικαιώματα επιμέλειας. Αυτό δεν ισχύει για τα δικαιώματα επίσκεψης. Και αν έχω δύο λεπτά μπορώ να δώσω το λόγο στη συνάδελφο, ίσως για τις απαντήσεις λέει η πρόεδρος. Γιατί πρέπει να ακούσουμε και τον άλλον προσύ... τον κύριο Μορτώνη. Εμένα η περίπτωσή μου δεν είναι ένας καυγάς γονιών για τα παιδιά όπως ε, συμβαίνει τακτικά. Απλώς ε, στις ε, γερμανικές αρχές δεν μπορώ, έχω το δικαίωμα να σκίσω το δικαίωμά μου ως πατέρας. Λοιπόν, η μητέρα του παιδιού με 500 χιλιόμετρα απόσταση μου επιβάλλει μία ψυχολογική πραγματογνωμοσύνη ότι δεν έχω δικαίωμα να συναντήσω το παιδί μου. Επίσης μου επιβάλλουν ε, την, την καταβολή διατροφής ενώ είμαι άνεργος στη Γερμανία και όλα αυτά με μια τεράστια χρονική καθυστέρηση. Μία επαγγελματίας η οποία επιλέγει από τη μητέρα λέει διάφορες ανακρίβειες χωρίς ημερομηνίε, χωρίς τίποτα ότι θα συναντήσω το γιο μου μόνο σε περίπτωση μόνο όταν θα πάει σχολείο διότι αυτό θα επιτρέπει στο γιο μου τον Μαξίμ να εκφράζει την επιθυμία του και τις ανάγκες του και θα μπορεί να απαντά λέγοντας όχι στις επιθυμίες του πατέρα. Το ναι δεν πάει καλά. Κανένας δεν θεωρεί ότι το να συναντήσω 16 ότι θα πρέπει μάλλον να συναντώ το παιδί μου 16 μήνων μία φορά κάθε 6 μήνες ε, συνοδευόμενο από μία babysitter η οποία, την οποία δεν είχε δει ποτέ του. Το παιδί ήταν ιδιαίτερα ευτυχισμένο όταν ήμουνα μαζί μου. Έκλαιγε μόνο όταν τελείωνε η συνάντησή μας. Κανένας δεν το δήλωσε αυτό. Λοιπόν, ζητώ εγώ από το γερμανικό δικαστήριο το δικαίωμα της διερμηνίας στο δικαστήριο. Λοιπόν, εγώ είμαι Ιταλός, δεν έζησα ποτέ στη Γερμανία, έπρεπε να ζήσουμε στην Ιταλία μαζί. Γνωρίζω πολύ καλά την Ιταλική γλώσσα και τη γνωρίζει και η μητέρα. Σήμερα για να δω εγώ το γιο μου πρέπει να μιλάω γερμανικά πρόκειται για παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Χάρτας. Ούτε με τον δίγλωσό μου δικηγόρο δεν μπορούσα εγώ να συναντήσω το παιδί. Και μία φορά έγινε αυτό υπό τον έλεγχο του Γιούγκενταλ. Και πρέπει να απαντώ εγώ μέσα σε τρεις εβδομάδες και στη δεύτερη ακρόαση το πρακτικό ήταν πάλι κατά εμού και δεν έχω το δικαίωμα καν της προσφυγής. Έχουν ένα, έχουν μία αρχή οι Γερμανοί δικηγόροι να εξυπηρετούν μόνο την γερμανική ένωμη τάξη και όχι τις αρχές της δικαιοσύνης και της ισότητας όπως τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Έτσι λοιπόν τελείωσε σήμερα όλη η διαδικασία αλλά δεν μου επιτρέπεται μια νέα ακρόαση γιατί το θεωρούν άχρηστο Παρότι ο γιος μου ο Μαξίμ, εδώ και ε, που είναι πια τεσσάρων ετών, πέφτει κάθε φορά στην αγκαλιά μου όταν με βρίσκει και εγώ δεν ξέρω πότε θα τον ξαναδώ. Του αφαίρεσαν και το επίθετό μου και δεν έχω την πατρική εξουσία. Θεωρώ λοιπόν ότι παραβιάζεται η σύμβαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών. Και ρωτώ λοιπόν γιατί η Γερμανία υπογράφει διεθνείς συμφωνίες και δεν τις στηρεί ποτέ και γιατί αφήνουμε σε αυτήν την χώρα το δικαίωμα του να προχωρεί σε διακρίσεις εκ μέρους της Κομισιόν. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να σας ενημερώσω για την αναφορά την οποία παρουσίασε η κυρία Κολόμπο. Όπως ακούσαμε, η αναφορά αυτή είναι πολύπλοκη. Υπάρχουν πολλές πτυχές που θα πρέπει να εξεταστούν. Καταρχάς, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πολύ προσεκτικά εξετάσει τις πτυχές αυτές και στην αναφορά προσπαθήσαμε να δούμε αν κάποιες από τις πτυχές της είχαν να κάνουν με την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου, της κοινοτικής νομοθεσίας. Καταρχάς θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να λάβει δράση μόνο σε περιπτώσεις παραβίασης θεμελιωδών δικαιωμάτων και όταν αυτά έχουν να κάνουν με την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, το ερώτημα το οποίο τέθη για την συμμετοχή της Jugendamt στην γερμανική διαδικασία, δικαστική διαδικασία, είναι μια διαδικασία που έχει να κάνει με το εθνικό δίκαιο και όχι με το κοινοτικό δίκαιο. Και γι' αυτό το λόγο δεν δύναται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθήσει περισσότερο το ζήτημα αυτό. Είναι καθαρά ζήτημα εθνικής δικαιοδοσίας. Όσον αφορά τα υπόλοιπα προβλήματα στα οποία αναφέρθηκαν οι ομιλητέ, θα ήθελα να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανακοίνωση που έκανε προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο λέει ότι ο περιορισμό τη ελεύθερη κυκλοφορία του αναφέροντος, αναφέροντος θα πρέπει να εξεταστεί ακόμα περισσότερο. Και γι' αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε τον αναφέροντα και ζήτησε από τον αναφέροντα πιο συγκεκριμένα να αποστείλει προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντίγραφα των συγκεκριμένων εγγράφων συγκεκριμένα τις αποφάσεις των Ιταλικών και Γερμανικών αρχών, έτσι ώστε να εξακριβωθεί περισσότερο το ζήτημα της αναλογικότητας και η έμπρακτη, ο έμπρακτος περιορισμός ελεύθερης κυκλοφορίας. Επίσης, η αναφέρουσα μας είχε πει ότι θα απέστελε τα έγγραφα αυτά πολύ σύντομα. Δυστυχώς, δεν έχουμε λάβει ακόμη εμείς τα έγγραφα αυτά. Και γι' αυτό το λόγο δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να αξιολογήσω την κατάσταση περαιτέρω. Θα ήθελα να καλέσω για άλλη μια φορά λοιπόν να φέρουσα να αποστείλει τα σχετικά έγγραφα, τα σχετικά αντίγραφα θέλετε των εγγράφων των δικαστικών αρχών, προκειμένου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταφέρει να δώσει μια απάντηση. Μετά την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η αναφέρουσα έδωσε κάποιες νέες απαντήσεις. Δυστυχώς και πάλι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είχε τον απαραίτητο χρόνο να εξετάσει περισσότερο τις απαντήσεις αυτές. Μόνο την προηγούμενη εβδομάδα καταφέραμε να τις μεταφράσουμε και γι' αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει μια νέα ανακοίνωση, ένα νέο έγγραφο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αργότερα. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει περισσότερο το ζήτημα της ε, εκείνης διαδικασίας Ιντερπόλ καθώς επίσης και τα άλλα ζητήματα στα οποία αναφερθήκατε. Αναφερθήκατε επίσης στην συνέχεια και στο ζήτημα της προάσπισης των συμφερόντων των παιδιών από τις γερμανικές αρχές. Ως προς αυτός πρέπει να σας πω ότι η αρχή της προάσπισης του συμφέροντος του παιδιού είναι μια πολύ σημαντική αρχή που συμπεριλαμβάνεται στην Σύμβαση των Εθνών για, για τα Δικαιώματα των Παιδιών, σύμβαση που έχει εγκριθεί, έχει επικυρωθεί από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να υπογραμμίσει ότι η εφαρμογή της κοινοτική νομοθεσίας θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με την αρχή αυτή. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι σε θέση να αξιολογήσει την εφαρμογή της αρχής αυτής σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Αυτό έχει να κάνει πάλι με την εθνική δικαιοδοσία, είναι, αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών. Επομένως δεν είμαστε σε θέση εμείς να αξιολογήσουμε ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή την εφαρμογή της αρχής της προάσπισης του συμφέροντος του παιδιού. Όσον αφορά τώρα την αναφορά του κυρίου Μολτόνη, θα ήθελα να σας πω ότι δεν έχει δοθεί ακόμα ανακοίνωση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ωστόσο θα μπορούσα εγώ να σας δώσω αυτή τη στιγμή κάποιες προκαταρχικές πληροφορίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί ότι το δικαίωμα σε μια δίκαιη δίκη, καθώς επίσης και το δικαίωμα της οικογενειακής ενότητας και το δικαίωμα μη διάκρισης είναι σημαντικές αρχές. Όπως είπα όμως και την περίπτωση της κυρίας Κολόμπο, Οι αρχές αυτές περιλαμβάνονται στην Χάρτα Θεμελιών Δικαιωμάτων, συγκεκριμένα στο άρθρο 51. Οι αρχές αυτές όμως έχουν να κάνουν με τις εθνικές νομοθεσίες και τους εθνικούς θεσμούς κάθε φορά που αυτοί εφαρμόζουν η κοινοτική νομοθεσία. Στην περίπτωση αυτή δεν μιλάμε για κοινοτική νομοθεσία αλλά για εθνική νομοθεσία, επομένως στην εθνική αρμοδιότητα. Η κυρία Γκρουνή έχει το λόγο. Δεν μπορώ να δώσω κάποια απάντηση αυτή τη στιγμή, παρόλα αυτά θα ήθελα να πάρω το λόγο. Θεωρώ ότι οι υποθέσεις αυτές είναι αρκετά δύσκολες βλέπουμε ότι εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε πολίτες δύο διαφορετικών κρατών μελών που αυτό συμβάλλει πολύ περισσότερο στην πολυπλοκότητα του ζητήματος αλλά ακόμα και στα πλαίσια ενός κράτους μέλους έχουμε αντίστοιχες περιπτώσεις. Στη Γαλλία για παράδειγμα ακόμα και όταν οι γονείς είναι και οι δύο Γάλλοι η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη και πολύπλοκη και στο όνομα κάθε φορά του συμφερόντος του παιδιού μπορεί και ο ένας και ο άλλος να υποβάλουν αρκετά θετικά επιχειρήματα. Ακούσαμε αυτή τη στιγμή, αν θέλετε, τη μία πλευρά μόνο του προβλήματος. Δεν έχουμε μπροστά μας συγκεκριμένα έγγραφα, δεν ακούσαμε την άλλη πλευρά. Αν κατάλαβα καλά, η κυρία Κολόμπο αναφέρθηκε σε γερμανική απόφαση και σε ιταλική απόφαση, οι οποίες αντιφάσκουν. Ε, όχι, όχι, δεν έχουν έτσι τα πράγματα. Η Ιταλική απόφαση, χωρίς μικρόφωνο. Στη μετάφραση τουλάχιστον που διάβασα εγώ κάτι τέτοιο λεγότανε ότι υπήρχε Ιταλική απόφαση υπέρ της κυρίας Κολόμπο, Γερμανική απόφαση κατά της κυρίας Κολόμπο. 9 Δεκεμβρίου το Ιταλικό Δικαστήριο ζήτησε τον επαναπατρισμό των δύο παιδιών στην Ιταλία. Αντίθετα, το Ιταλικό Δικαστήριο ζήτησε επαναπατρισμό στη Γερμανία και ε, το εφετείο επικύρωσε την απόφαση. Ο Άριος Φάγος. Λοιπόν, αλλά μετά να ξαναμιλήσετε. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, είναι πολύ δύσκολο για μας αυτή τη στιγμή να τοποθετηθούμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την άλλη δεν έχει το σύνολο των απαραίτητων εγγράφων που θα μας επέτρεπαν να βοηθήσουμε τους αναφέροντες. Σε κάθε περίπτωση πάντως το ζήτημα του συμφέροντος του παιδιού είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό, για μένα κάτι το θεμελιώδες πριν από λίγο ακούσαμε ότι στην Γαλλία υπήρχε ένα συνήγορος του παιδιού και του εφήβου που δεν υφίσταται πλέον. Ουσιαστικά τον ρόλο του συνηγόρου του παιδιού έχει αναλάβει ο συνήγορος του πολίτη. Και αυτό είναι πραγματικά κρίμα, γιατί θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε έναν θεσμό ουδέτερο που θα μπορούσε να τοποθετείται υπέρ του συμφέροντος του παιδιού. Στην Γαλλία τα γαλλικά δικαστήρια καλούνται πολύ συχνά να εκδικάσουν τέτοιε υποθέσει, οι οποίε είναι πάρα πολύ δύσκολε. Εμεί, τουλάχιστον στη δικιά μου περιοχή στη Γαλλία, προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε μια αρχή διαμεσολάβηση, η οποία θα μπορούσε να διευκολύνει την εξέταση τέτοιων υποθέσεων, οι οποίε πάντα παρεμένουν πολύ δύσκολε βέβαια. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θυμάμαι στην προηγούμενη θητεία είχαμε ακριβώς για αυτό το θέμα του Jugendamt πάρα πολλές αναφορές και πάρα πολλές συζητήσεις. Θα το θυμούνται οι παρόντες. Ε, δεν ήταν μόνο Ιταλοί, ήταν και από την Πολωνία νομίζω, αν θυμάμαι καλά, τα παιδιά. Και η συζήτηση αρκετά θερμή και με ε, πολλά πάθη για την κατάσταση αυτή. Εγώ δεν θέλω να μπω στην ουσία των όσων είπε η κυρία Γκρουνή, γιατί τα εξήγησε πάρα πολύ καλά, αλλά θα ήθελα μόνο σε σχέση με τα όσα είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και απάντησε και για να δώσουμε λίγο φως αυτή τη συζήτηση για να μην φύγουν οι αναφερόμενοι χωρίς απάντηση νομίζω ανοίγει μια πόρτα εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους εκπροσώπους του Κοινοβουλίου επίσης. Λέει και η Κομισιόν ότι περιμένει λεπτομέρειες για τις δικαστικές αποφάσεις για να μπορέσει να τις εξετάσει. Θα μπορούσαμε λοιπόν να ζητήσουμε από τους ενδιαφερομένους, τους αναφερομένους περισσότερα στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προτείνω αυτή η αναφορά να μην κλείσει, να παραμείνει ανοιχτή και με ε, αυτά που ζητάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ενημέρωση που θα στείλουν οι ενδιαφερόμενοι η αναφερόμενη προκειμένου να ε, διευκρινιστεί αυτό το θέμα, να γνωρίζει περισσότερα στοιχεία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να λυθεί το πρόβλημα, γιατί αυτό που θέλουμε τελικά είναι να δώσουμε διέξοδο και να ε, δικαιωθούν οι άνθρωποι να έχουν μια σαφή, ε, συγκεκριμένη απάντηση του Κοινοβουλίου και συνεκτική και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν συμφωνείτε κυρία Πρόεδρε, να μην κλείσουμε και αν συμφωνούν και αναφερόμενοι βεβαίως. Κολέγα ο Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω τη γλώσσα μου. Τρεις παρατηρήσεις θα ήθελα να κάνω. Πρώτον, Όταν βλέπουμε ότι δεν εφαρμόζεται σωστά η νομοθεσία, είτε πρόκειται για τη γερμανική νομοθεσία, την ιταλική, τη ρουμανική νομοθεσία, σε κάθε περίπτωση οι υποθέσει αυτέ θα πρέπει να αποτελούν αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και θα πρέπει να διευκρινίζονται πολύ περισσότερο οι σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών, δηλαδή να διευκρινίζεται πολύ περισσότερο η αρχή τη επικουρικότητα. Όταν έχουμε πολίτε οι οποίοι είναι θύματα αποφάσεων που ουσιαστικά αντιτίθενται στην εθνική νομοθεσία ενός κράτους μέλους, τότε οι πολίτες αυτοί θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και θα πρέπει να λαμβάνουν και αποζημίωση. Επίσης εκπλήσω που βλέπω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ιδιαίτερα ασαφής όσον αφορά τον χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Από όσο γνωρίζω εγώ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επικυρώσει το χάρτη αυτό Και αυτό έχουν πράξει άλλωστε και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή τη στιγμή λοιπόν επικυρώνεται ένα τέτοιο χάρτη, όπω ο χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων, αυτόματα η εφαρμογή του εγγράφου, που αποτελεί πλέον νομικό έγγραφο, θα πρέπει να εξασφαλίζεται. Καταλαβαίνετε ότι δεν ήταν ένα τυχαίο έγγραφο, ένα έγγραφο μιας κάποιας δεοντολογίας που έπρεπε να ακολουθηθεί. Πρόκειται για ένα νομικό έγγραφο, πρόκειται για νόμο πλέον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έρχεται και μας λέει ότι κάποια τμήματα του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων μπορούν να εφαρμοστούν στα κράτη-μέλη και ότι έχουν νομική ισχύ, ενώ υπάρχουν και κάποια άλλα τμήματα του χάρτη που δεν έχουν νομική ισχύ, που δεν έχουν εισάξει νομική ισχύ τουλάχιστον. Αυτό φαίνεται να μας λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ζήτημα αυτό θα ήθελα να το θίξω στην κυρία Ρέντινγκ όταν θα έρθει σήμερα το απόγευμα. Νομίζω ότι θα πρέπει συντομότατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσει την κατάσταση και να μας πει πώς εφαρμόζεται ή πώς δεν εφαρμόζεται ο χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Γιατί αν δεν διευκρινιστεί η κατάσταση, τα πράγματα παραμένουν πάρα πάρα πολύ ασαφή και οι Ευρωπαίοι πολίτες θα έρχονται εδώ στην Επιτροπή μας και θα ανακαλύπτουν ότι δεν μπορούμε εμείς να τους βοηθήσουμε ακόμα και όταν έχουν δίκιο. Πρέπει λοιπόν να ξεκαθαριστεί το ζήτημα αυτό θα πρέπει να αποσαφινιστεί το ζήτημα το συντομότερο δυνατό. Σας ευχαριστώ. Äh, λοιπόν, αν κατάλαβα καλά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι μας λέει. Ότι δεν είναι σε θέση ε, να κρίνει τα θέματα που μας ενδιαφέρουν εμάς. Γιατί τις λείπουν πολλά στοιχεία. Ε, ας αφήσουμε ανοιχτή την αναφορά, εντάξει. Αλλά την άλλη φορά να μα απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όχι να ξανάρθουμε την άλλη φορά και να μα πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ξέρετε μου λείπουν κάτι πληροφορίε ακόμα. Και κάτι άλλο που περιπλέκει τα πράγματα, Έκανα την εξή ερώτηση προηγουμένω και στο, για την κυρία Κολόμπο. Για τη δικαιοδοσία και για την αναγνώριση. Ορίστε, ειδού έχουμε μια απόφαση δικαστική γερμανικού δικαστηρίου και ο αναφερόμενο τότε δεν έκανε έφεση ε, για ε, ε, την απόφαση αυτή, οπότε και είναι έγκυρη πλέον νομικά. Δεν το ξέχασε ή έχασε τις προθεσμίες ή δεν θέλει, σε περιπτώσει τώρα αυτό είναι τελικό. Και άκουσα καλά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μας λέει ότι δεν μπορεί ακόμα να αποφανθεί οριστικά παρόλο μάλλον εάν παραβιάζεται κοινοτικό δίκαιο οι αποφάσεις Εντάξει, τις λείπουν πληροφορίες, αλλά την άλλη φορά παρακαλώ να ξαναμπεί η αναφορά στην ημερήσια διάταξη μόνο και, ε, τότε και μόνο τότε όταν έχει ε, τις πληροφορίες στη διάθεση τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διότι ξέρουμε ότι υπάρχουν τα δικαιώματα του πατρός, της Μητρό, αλλά κυρίω του παιδιού. Αυτό είναι το μαγικό τρίγωνο φυσικά, δούμε πώ θα μπορέσουμε να το λύσουμε, το τετραγωνισμό του κύκλου. Και το Jugendamt στη Γερμανία, ε, ακριβώς γι' αυτό το λόγο δημιουργήθηκε αυτός ο θεσμός, για να εκπροσωπεί το συμφέρον του παιδιού. Όταν διαπληκτίζονται ο πατέρας και η μητέρα, ε, αυτός ο οργανισμός που ε, ασχολείται με την νεολαία ε, αυτεπάγγελτα επεμβαίνει για να διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού από την ίδια τη φύση του και τη, τη, του και τη λειτουργία του το Jugendamt Jugendamt. Κάθε χώρα το βλέπει διαφορετικά το πράγμα. Στη Γερμανία λέγεται έτσι αυτός ο οργανισμός. Παράδειγμα, το παιδί μου. Ε, ας πούμε στο δικό μου οικόπεδο πέρασε απέναντι δίσχυσε ένα δρόμο που απαγορευόταν η, διάβαση των πεζών και ε, αυτό είναι ε, παράβαση του νόμου. Ε, ε, ε επενεύει ωστόσο, παρόλα αυτά που ήταν ξεκάθαρη περίπτωση, επενεύει το Jugendamt για να δει τι γίνεται στο σπίτι μου, τι κατάσταση επικρατεί, πώς είναι το παιδί και τι περνάει. Και δεν έχει καμία σχέση με διακρίσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Αχ, συγγνώμη, ήθελα να τονίσω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, εντάξει, διαπληκτίζονται οι, οι γονείς, γι' αυτό απευθύνονται σε δικαστήρια. Αλλά το παιδί ποτέ τον ποτέ τον ποτόν, ουδέποτε δεν θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο της διαφωνίας και της ε, διέναξης των γονέων. Να μην τσακώνονται για το παιδί. Γι' αυτό χρειαζόμαστε αυτό το Jugendamt, αυτή την υπηρεσία που έχει ως ύψιστο αγαθό την ευημερία και το συμφέρον και το ενδιαφέρον του παιδιού. Και θέλουν ε, τα δικαστήρια να βοηθούν το παιδί. Οι γονεί δεν έχουν αξίωση ε, στα, ε, επί των παιδιών του, δεν έχουν δικαιώματα στα παιδιά του. Το παιδί έχει δικαίωμα σε μια ευημερούσα και αξιοπρεπή ζωή. Ευχαριστώ. Λοιπόν, εγώ το πρώτο πράγμα που ρωτώ σε εσά είναι πώ το Jugendamt διαφύλαξε τα συμφέροντα του παιδιού που το βασικό του δικαίωμα είναι να έχει δυο γονείς αποκλείοντας τη μαμά για δέκα μήνες χωρίς καν να μπορεί να τηλεφωνήσει. Αν μου το πείτε εσείς που διαφυλάσσετε αυτό, εξηγήστε το μου και εγώ μετά δεν λέω πια τίποτα. No, però non, non so. Συγγνώμη, εγώ δεν μπορώ να δώσω το λόγο σε όλους για αυτό το θέμα. Μου ζητήσατε... Είμαι η δικηγόρος ε, Κουντέρη και εκπροσωπώ την κυρία Κολόμπο. Λοιπόν, παρακαλώ να είστε σύντομοι. Διότι η αναφορά θα μείνει ανοιχτή κατόπιν αιτήματος των όλων θα πρέπει να δώσουμε πιο σαφή εντολή στην Κομισιόν για να απαντήσει. Το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών ορίζεται στην απόφαση που επιβάλλει στην κυρία Κολόμπο να μην πάει με τα παιδιά της στην Ιταλία. Λέει ότι η ελεύθερη κυκλοφορία της μητέρας ε, δεν θα πρέπει να ε, εμποδίζει το δικαίωμα επαφής του πατέρα με τα παιδιά. Εσείς πιστεύετε ότι εδώ εγγυάται κανείς την ελεύθερη κυκλοφορία των ε, παιδιών ή διακρίσεις που έχουν να κάνουν και με την υπηκότητα των πολιτών για το Jugendamt δεν αφορούν το κοινοτικό δίκαιο δεν αφορούν με τίποτα το αντικείμενο της Κομισιόν με το οποίο θα μπορούσε να ασχοληθεί. Ευχαριστώ. Εσείς δεν έχετε υπογράψει την αναφορά, οπότε κλείνω το θέμα. Σχετικά λοιπόν με αυτήν την αναφορά θα προσέθετα το εξής προς την Κομισιόν. Όταν θα αρχίσει να ελέγχει τα έγγραφα που ο εκπρόσωπος της αναφοράς για την κυρία Κολόμπο θα καταθέσει για να εμβαθύνετε στην αξιολόγησή σας που είναι η αρχή δηλαδή της παραβίασης της οδηγίας κατά των διακρίσεων που αποτελεί τμήμα του ευρωπαϊκού δικαίου που θέτουν ε, ως επιχείρημα οι συντάκτες της γνωμοδότησης, ας πούμε η απόλυτη γνώση της γερμανικής γλώσσας. Αυτό δεν παραβιάζει την ελεύθερη κυκλοφορία ε, των πολιτών και την, και ισοτιμία των κρατών μελών και των γλωσσών τους και τη χρήση τους στις 27 χώρες. Η αναφορά παραμένει ανοιχτή με όλες τις παρατηρήσεις και θα αποφασίσουμε έγκαιρα με περισσότερες διευκρινήσεις από την Κομισιόν. Επόμενο σημείο. 9. Ο κύριος Έλβιο Γκάλο. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Αξιοσέβαστη Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Συνθήκη λέει ότι εμπνέεται από τις θεμελιώδεις ελευθερίες του ανθρώπου και θεωρεί ότι είναι απαραβίαστες. Ο άνθρωπος έχει δικαιώματα που του ανήκουν από το φυσικό δίκαιο και τα κράτη δεσμεύθηκαν με την επικύρωση των συνθήκων να αναγνωρίζουν αυτά τα δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας το Δεκέμβριο του 2009 η χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων έχει την ίδια νομική αξία με τις συνθήκες. Έτσι λοιπόν τονίζεται ακόμη περισσότερο ο ρόλος του ατόμου ως πρόσωπο και τονίζεται το πρόσωπο με έμφαση, δηλαδή δίνοντας στον πολίτη ένα πιο κεντρικό ρόλο. Η συνθήκη στα άρθρα 2 και 3 ε, καλεί στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στα δικαιώματα των ανηλίκων και στο άρθρο 4 ζητάν την ε, νόμιμη συνεργασία και στο άρθρο 5 ορίζει τις ε, αρχές αρμοδιότητας, ε, επικουρικότητας και αναλογικότητας. Εγώ, όσα μάλλον ορίζονται στο άρθρο 2 ενισχύονται στο άρθρο 7. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως φρουρός των συνθήκων έχει σημαντικό ρόλο στην ε, διαφύλαξη των δικαιωμάτων της χάρτας. Στο άρθρο 1 λοιπόν της χάρτας ε, τονίζεται η περιφρούνηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και εμένα έχει καπατηθεί η αξιοπρέπειά μου αρνήθηκαν να με ενημερώσουν για το πώς εξελίσσεται η εγκυμοσύνη και μου στέρισαν το δικαίωμα να είμαι παρόν κατά τη γέννηση του γιού μου. Δεν μπόρεσα εγώ ακόμη σήμερα να γνωρίσω το γιο μου. Στο άρθρο 2 που αφορά ελευθερία λέει το, αναφέρεται το άρθρο 7 το οποίο επικαλείται το άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου σχετικά με την ιδιωτική και την οικογενειακή ζωή. Στον τρίτο τίτλο αναφέρεται το άρθρο 20 και λέει ισονομία 21, μη διάκριση, 23, ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Άρθρο 24, δικαιώματα του ανηλίκου όσον με αφορά. Τα πρώτα τρία άρθρα, άμα τα συνδυάσουμε μαζί, ε, ε καθιστούν καταφανές πως εγώ και λόγου φίλου στην διακρίση στην προσπατασία των δικαιωμάτων μου και οδηγήθηκα και σε, δαπανι, σε τεράστιες νομικές δαπάνες και αυτό επιβαρύνει και το παιδί μου το οποίο ορίζεται ως τέκνο αγνώστου πατρός και του αρνούνται το δικαίωμα να γνωρίσει τον πατέρα του. Οι σχετικές αρχές και δικαστήρια έχουν ενημερωθεί. Στο άρθρο 24 που έχει ως τίτλο «Δικαιώματα του παιδιού» πώς ε, αντιπροσωπεύεται σε επίπεδο δικαιοδοσιών, στο άρθρο 45 λέγεται ότι η ελευθερία της ελευθερίας και διαμονής είναι ένα δικαίωμα το οποίο δεσμεύεται από τις συνθήκες η κατάχρηση της ε, μητέρας που επανήλθε στη Γαλλία, επέστρεψε στη Γαλλία στον τέταρτο μήνα της εγκυμοσύνης εκμεταλλεύτηκε τα πολιτικά και νομικά εμπόδια εμποδίζοντάς μου να ασκήσω τα δικαιώματά μου. Υπάρχουν ε, σήμερα εμπόδια μεταξύ Γαλλίας, ε, στην και... μεταξύ Γαλλίας και Ιταλίας που παρεμποδίζουν την αναγνώριση των δικαιωμάτων μου ως Ευρωπαίου πολίτη. Θεωρώ ότι αυτή η έλλειψη αναγνώρισης των δικαιοδοσιών και συνεργασίας των δικαιοδοσιών βρίσκονται στη βάση της καταπάτησης των δικών μου δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων του παιδιού μου. Μετά άρθρα 51, 52 και 54 πρέπει να ορίσουμε ως κατάχρηση δικαιωμάτων εκείνη την παρανομία που στοχεύει στην καταστροφή των δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται από την παρούσα χάρτα. Εγώ τρέφω εμπιστοσύνη στην υλοποίηση μιας καλύτερης Ευρώπης γιατί ως πατέρας εύχομαι στο, στο γιο μου να μπορέσουμε να εγγυθούμε μια ε, ζωή όσο το δυνατόν πιο ήρεμη. Σας ευχαριστώ πολύ. Μυριάμ Ντεμίχ από την Κομισιόν. Δεν είναι εδώ. Είναι. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ κύριε Γκάλο που παρουσιάσατε την αφορά σας αυτή. Θα ήθελα να σας πω καταρχάς ότι η αναφορά αυτή θέτει πάρα πολλά ερωτήματα και πάρα πολλά ζητήματα. Το ζήτημα της σχέσης, της συγγένειας, συγκεκριμένα αναφερόμαστε εδώ πέρα στον πατέρα και αναφερόμαστε επίσης και στο ζήτημα της νομικής βάσης όσον αφορά την θέσπιση του δικαιώματος συγγένειας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε υπόψη της όλα τα ζητήματα τα οποία θέτει αναφορά του κ. Γκάλου Μέχρι στιγμής το ζήτημα της αναγνώρισης της συγγένειας δεν αποτελεί αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά αρμοδιότητα των κρατών μελών. Αποτελεί δηλαδή αντικείμενο της εθνικής νομοθεσίας. Ο κανονισμός Βρυξέλλες 2 της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν καλύπτει το ζήτημα της συγγένειας. Επομένως, είναι η εθνική νομοθεσία αυτή η πλέον αρμόδια για να αποφανθεί για το ζήτημα το οποίο θέτει ο κύριος Γκάλο. Συνεπώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι σε θέση να συμβάλλει περισσότερο και δυστυχώς το μόνο το οποίο μπορεί να ζητήσει είναι να κλείσει η αναφορά αυτή. Ωστόσο, θα ήθελα να απογραμμίσω ότι μέσω της αναφοράς αυτής η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να αναφερθεί στις πάρα πολλές δυσκολίε που παρουσιάζονται αυτή τη στιγμή σε ζητήματα αστικών υποθέσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργάζεται αυτή τη στιγμή ε, μία πράσινη βίβλο για την αναγνώριση των αποφάσεων σε αστικές υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προτίθεται να ξεκινήσει μία ευρεία διαβούλευση η οποία πιστεύω θα μας δώσει την δυνατότητα να εφαρμόζεται περισσότερο και να αναγνωρίζονται οι αποφάσεις σε αστικές υποθέσεις παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ. Επιθυμεί κάποιος συνάδελφος να πάρει το λόγο. Κυρία Γκρούνη, σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και στην περίπτωση αυτή θα έλεγα ότι δεν μπορούμε να δώσουμε μια κάποια συγκεκριμένη απάντηση και αυτό γιατί στην Γαλλία τουλάχιστον δεν έχουμε βρει ακόμα μια απάντηση για το ερώτημα αυτό. Ξέρω πολλές νέες γυναίκες οι οποίες αποκτούν τα παιδιά τους μόνες τους. Οι πατέρες πολλές φορές δεν το γνωρίζουν ή ακόμα και το γνωρίζουν δεν έχουν αναγνωριστεί. Καταλαβαίνω λοιπόν πολύ την απόγνωση που νιώθει ο Κύριος εδώ. Δυστυχώς όμως δεν μπορούμε να πούμε εμεί τώρα τίποτα παραπάνω. Σαφώς καταλαβαίνουμε τις ανησυχίες σας, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να σας δώσουμε μία νομική απάντηση. Δεν νομίζω λοιπόν ότι θα ήταν χρήσιμο ακόμα και να αφήνουμε την αφορά αυτή ανοιχτή. Δυστυχώς δεν μπορώ να σας πω τίποτα παραπάνω. Πραγματικά, ειλικρινά, λυπάμαι. Θέλει κανείς άλλος να στο λόγο. Η κυρία Όκεν, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να συμφωνήσω απολύτως με την κυρία Γκρινή. Τι γνωρίζουμε αυτές τις ιστορίες από όλα τα κράτη μας, για να μην πω και από τις ίδιε μα οικογένειε. Και πολλές φορές ε, είναι πολύ τραγικό αυτό και πολύ εκνευριστικό, αλλά οι αρχές ε, ε, στα διάφορα κράτη-μέλη προσπαθούν να προστατεύσουν τα παιδιά να μην γίνουν το αντικείμενο της έρηδος των γονέων τους αυτό που ενδιαφέρει είναι αποκλειστικά το ε, συμφέρον και το ενδιαφέρον του παιδιού. Ακόμα και αν αδικείται κάποιος από τους γονείς. Δεν είναι αυτό το πρίσμα και θα πρέπει να σεβαστούμε αυτό το πρίσμα ότι αυτό που προέχει και είναι αποφασιστικό είναι τα δικαιώματα των παιδιών και όχι των γονέων ε, ενό εκ των δύο εν πάση περιπτώσει. Και παρακαλώ να κλείσει εδώ αυτή η αναφορά. Ο κύριος ε, Κυρία Πρόεδρε, έχω την άποψη ότι σε αυτή την ειδική περίπτωση πρόκειται απολύτως περί του δικαιώματος του παιδιού. Ένα αυτό. Δεύτερον, είναι θέμα επικορικότητας. Και αν υπάρχουν προβλήματα που συνδέονται με τα δικαιώματα του πατρός, της μητρός ή της υποχρεώσεις ή της δεσμεύσης, αν είναι θέμα αστικού δικαίου, τότε αυτό θα πρέπει να πάει σε ένα αστικό δικαστήριο, το οποίο ενδεχομένως να είναι αρμόδιο, να το εξτάσει και τελικά να δοθεί κάποια απάντηση στον αναφερόμενο. Τελεία. Οπότε και εγώ είμαι υπέρ του να κλείσει εδώ αυτή η αναφορά. Και να προχωρήσουμε και πάλι κάτι που είναι δική μου αιμονή. Θα πρέπει να αποφεύγουμε τις δυνατότητες της όσο γίνεται να μην επεμβαίνουμε σε θέματα που δεν αφορούν ε, άμεσα ευρωπαϊκούς κανόνες. Ξέρω ότι είναι ευαίσθητο το θέμα, τα δικαιώματα των γονέων, το καταλαβαίνω. Πάντα είναι πολύ σημαντικά αυτά, αλλά προκειμένου θα ζητούσα κι εγώ να κλείσει ένα φορά. Όπως πρότεινε η κυρία Γκρίνη. Ευχαριστώ. Υπάρχει σαφής πλειοψηφία. Εμένα με, με καθιστά αμήφανη η σοβαρότητα του θέματος, αλλά χρειάζεται να υποκύψω στη βούληση των συναδέλφων που λένε ότι δεν είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής μας σχετικά. Επιτρέψτε μου απλώς μία παρατήρηση σχετικά με τη δική μας προτεραιότητα που είναι να προστατεύσουμε τα συμφέροντα των ανηλίκων και όχι των παιδιών και όχι των ε, γονέων, συγγνώμη. Εμείς είμαστε πεπισμένοι από όλα όσα ακούμε και όσα γεγονότα μας αναφέρονται εδώ δεν έχουμε παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανηλίκου. Ε, ε, μένοντας λοιπόν στη Γενική Αρχή Θα το συζητήσουμε και με τους συντονιστές. για να ξανασυζητήσουμε το θέμα, όχι όντας εμείς δικαστές, γιατί δεν είμαστε δικαστές, ούτε υποκαθιστούμε το εθνικό δίκαιο. Απλώς θέλουμε να προστατεύσουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα τα οποία εμπνέουν το ευρωπαϊκό δίκαιο. Λοιπόν, το σημείο 13 ζητήθηκε να το εξετάσουμε πριν από το σημείο 10 διότι ο εκπρόσωπος της Κομισιόν πρέπει να φύγει από την αίθουσα. όντας παρόν ο εισηγητής ε, ο κύριος Μάρτιν Καρμπόφσκι για την ε, αναφορά 099 2008 δίνω το λόγο στον ε, κύριο Αλόνσο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ που λάβατε υπόψη στο έτοιμά μου. Έχουμε εδώ πέρα μία αναφορά που έχει να κάνει με μία πολύ σοβαρή περίπτωση στη Βουλγαρία, όπου λέγεται ότι παιδιά και παιδιά τα οποία βρίσκονται κυρίως σε ιδρύματα έχουν πέσει θύματα σεξουαλικής κακοποίησης. Και η απόφαση ουσιαστικά όλων των δικαστηρίων που έχουν ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό είναι η ατιμορρησία. Ατιμορρησία για αυτούς που κατηγορούνται για την παιδοφιλία, για την κακοποίηση, που είναι πολύ συχνά άνθρωποι που βρίσκονται σε πολύ υψηλέ διοικητικέ θέσει. Καταλαβαίνετε ότι μα αναστατώνει πάρα πολύ το ζήτημα αυτό, είναι πάρα πολύ σοβαρό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται για την καταπολέμηση των ιδεχθών αυτών εγκλημάτων, εγκλήματα τα οποία δημιουργούν ανεξίτηλα ίχνη τραύματα στα παιδιά. Λαμβάνοντα λοιπόν τα δεδομένα αυτά υπόψη, θα πρέπει να αναρωτηθούμε τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το πρόβλημα. Αυτό το οποίο δεν μπορούμε να κάνουμε είναι να αναθεωρήσουμε δικαστικές αποφάσεις που έχουν ληφθεί σε εθνικό επίπεδο, στα πλαίσια της ποινική διαδικασίας. Αυτό σαφώς δεν μπορεί να γίνει. Αυτό που μας ανησυχεί όμως σε συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι φαίνεται να υπάρχει μία γενικότερη τάση για κάποιες συγκεκριμένε πολιτικές και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δει πώς αυτές οι εθνικές πολιτικές που βλέπουμε να δίονται έρχονται σε αντίθεση με κάποια ευρωπαϊκά πρότυπα. Υπάρχουν κάποια ευρωπαϊκά πρότυπα τα οποία θα μπορούσαν να προστατεύουν τα παιδιά από την σεξουαλική εκμετάλλευση. Τα πρότυπα θα πρέπει να τα αποκρίνονται σε δύο κριτήρια. Πρώτον, να δίνουν απαραίτητη προστασία στα παιδιά. Θα πρέπει προφανώ να μιλάμε για υψηλά κριτήρια, υψηλά πρότυπα, τα οποία να εγγυώνται αυτή την ασφάλεια, αυτή την προστασία. Και τα ευρωπαϊκά πρότυπα θα πρέπει να είναι σαφώ δεσμευτικά, ώστε τα κράτη-μέλη να μην μπορούν να τα παρακάμψουν. Έχουμε εμεί τέτοια πρότυπα αυτή τη στιγμή. Η απάντηση είναι όχι. Δεν έχουμε τέτοια πρότυπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε κοινοτική νομοθεσία έχουμε συγκεκριμένα μια απόφαση πλαίσιο η οποία έχει ως στόχο να προσεγγίσει περισσότερο την εθνική νομοθεσία. Το 2004 υπάρχει απόφαση αυτή, η οποία δυστυχώς περιλαμβάνει τα ελάχιστα κριτήρια προστασίας και τα ελάχιστα αυτά κριτήρια είναι αρκετά χαμηλά τελικά. Αναφέρεται μόνο σε κάποια πάρα πολύ σοβαρά εγκλήματα και ζητά από τα κράτη-μέλη να ποινικοποιούν τα εγκλήματα αυτά, αλλά το επίπεδο για παράδειγμα των κυρώσεων δεν μπορεί να είναι αποδεκτό. Για παράδειγμα, σύμφωνα με αυτό το σύμφωνο πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση ικανοποιείται με μία μέγιστη ποινή τριών ετών. Για τις πιο σοβαρές μάλιστα υποθέσεις, η μέγιστη ποινή προβλέπεται από την απόφαση πλαίσιο θα μπορούσε να είναι πέντε χρόνια. Μιλάμε για μέγιστη ποινή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η πραγματική ποινή θα είναι πάντα χαμηλότερη το υφιστάμενο επίπεδο προστασίας σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά κριτήρια δεν είναι αυτό το οποίο αναμένουν από εμά οι Ευρωπαίοι πολίτες. Πρώτον αυτόν. Δεύτερον, τα κριτήρια αυτά πολύ δύσκολα μπορούν να εφαρμοστούν. Και αυτό γιατί τα κράτη-μέλη πρέπει να εγκρίνουν σαφώ νομοθεσία, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο εναντίον των κρατών μελών για τα ζητήματα αυτά. Δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο από τη συνθήκη. Συνεπώς χρειαζόμαστε τα κριτήρια αυτά στα οποία αναφέρθηκα και θα πρέπει τα κριτήρια, τα πρότυπα με να ανταποκρίνονται σε αυτά τα δύο κριτήρια. Και αυτό προσπάθησε να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Μάρτιο του 2010 Λίγου μήνε μετά τη θέση εφαρμογή της συνθήκης Λισαβόνα, Υποβάλαμε συγκεκριμένα πρόταση για μια οδηγία η οποία θα καταπολεμεί την κακοποίηση των παιδιών, τη σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών, την κακομεταχείριση και την παιδοφιλία, καθώ επίση και την παιδική πορνογραφία. Πρόκειται για μια πρόταση την οποία θα πρέπει να εξετάσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και σύμφωνα με την απόφαση αυτή μπορεί να οδηγηθεί στο δικαστήριο ο υπεύθυνος το επίπεδο προστασίας που ζητείται εδώ πέρα είναι πολύ πιο υψηλό. Θέλουμε να αυξηθούν επίσης οι κυρώσεις, το επίπεδο των κυρώσεων. Θα πρέπει η ποινή να είναι αναλογική, αποτελεσματική και να είναι και αποτρεπτική. και θα πρέπει να περιοριστεί πολύ σημαντικά το περιθώριο τιμωρησία. Πρόκειται λοιπόν για μια πολύ σημαντική πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δεν έχει να κάνει μόνο με την προσφυγή κατά του ε, ένοχου, αλλά δίνει τη δυνατότητα και στις ε, εθνικές αρχές να αναλάβουν την απαραίτητη δράση προκειμένου να σταματήσουν εγκληματία. Προβλέπονται επίσης ε, κανόνες που θα μπορούσαν να σταματήσουν τον εγκληματία, τον ένοχο, από το να πηγαίνει σε μία άλλη χώρα προκειμένου να αποφύγει την ε, ποινή. Προβλέπεται επίσης προστασία του θύματος, το οποίο ήδη έχει περάσει μια τραυματική εμπειρία και δεν θα πρέπει η εμπειρία του αυτή να επιδεινωθεί μέσω της δικαστικής διαδικασίας. Έχετε μπροστά σας λοιπόν εσείς την πρόταση αυτή, την πρόταση θα εξετάσει και το Συμβούλιο. Σαφώς πρέπει να γίνουν περισσότερα πράγματα. Όσον αφορά όμως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η βασική πρόταση αυτή τη στιγμή έχει υποβληθεί. Θεωρούμε λοιπόν ότι εναπόκειται πλέον στα άλλα δύο θεσμικά όργανα, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Συμβούλιο, να λάβουν δράση και να εγκρίνουν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βρίσκονται σε εξέλιξη οι συζητήσεις και ελπίζουμε ότι την δέσμευση που, δίνει, που δείχνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα τη δείξουν και τα άλλα δύο θεσμικά όργανα. Είμαι βέβαιος αστικά γι' αυτό. Ελπίζω ότι μετά από όλα αυτά μπορεί να κλείσει η συγκεκριμένη αναφορά. Ευχαριστώ. Θέλει κανεί το λόγο. Μποστινάρου. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, την περασμένη άνοιξη το Κοινοβούλιο με συντριπτική πλειοψηφία ενέκρινε μια διακήρυξη για την καταπολέμηση ε, της ε, ε, σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών και της πορνογραφίας και της παιδεραστίας ή παιδοφιλίας. Ε, θα ρίνομαι πάρα πολύ από αυτά που μας λέει σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είμαι πεπισμένος επίσης ότι προσεχώς το σχέδιο αυτό θα καταστεί ένα νομικά δεσμευτικό μέσο για όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης. Μπορεί να υπάρχουν και πολιτικά και προσωπικά συμφέροντα στο μεταξύ για να μην είναι τόσο σκληροί οι κανόνες. Θα πρέπει όμως να κάνουμε ό,τι μπορούμε, να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να περάσει η πιο αυστηρή λύση, η πιο σκληρή λύση για την καταπολέμηση, επαναλαμβάνω αυτών των καταστάσεων της σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών, της κακομεταχείρισης και της παιδεραστίας. Γιατί χρειαζόμαστε ένα πανευρωπαϊκά ε, δεσμευτικό νομικό εργαλείο. Γιατί είναι τραγική η κατάσταση, όχι μόνο στη Βουλγαρία, όπως ανέφερε ο αναφερόμενος, αλλά και στη δική μου χώρα. Και δεν είναι μόνο οι πολίτες των κρατών αυτών, αλλά και πολλοί άλλοι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενέχονται και πολλές φορές μέσω των νομικών διατάξεων που ισχύουν ε, ανά περίπτωση καταφέρνουν να ε, επιτυχάνουν ε, λιγότερο αυστηρή δικαστική απόφαση από ό,τι στις δικές τους χώρες. Ή από ό,τι αν το δίκαζε αυτά ένα ε, βουλγαρικό ή ένα ρουμανικό δικαστήριο. Και είμαι πεπισμένος ότι η μοναδική λύση εδώ είναι μια ε, νομική, νομικά δεσμευτική συγγνώμη, λύση σε όλη την Ένωση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω μόνο ότι είναι καλό, είναι θετικό που είναι υπό παρακολούθηση η κατάσταση αυτή στη Βουλγαρία σε θέμα δικαιοσύνης και εσωτερικών και μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακριβώς να παρακολουθεί ε, τα τεκτενόμενα στη χώρα. Γίνεται λόγος για ένα ευρωπαϊκό νομικό εργαλείο. Μα κύριε Μποστινάρου υπάρχουν ήδη τέτοια στοιχεία συνεργασία και καμιά φορά το πρόβλημα είναι ότι ε, υπάρχουν και νόμοι και θεσμοί, αλλά δεν τηρούνται, δεν εφαρμόζονται και οι θεσμοί δεν εργάζονται αποτελεσματικά. Γι' αυτό στην περίπτωση αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύω ότι έχει μέσα να επέμβει με αυτό το σύστημα παρακολούθησης, αν θέλετε, ε, της Βουλγαρίας σε θέματα δικαιοσύνης και εσωτερικών. Η κυρία Γιώτοβα, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να προτείνω η αναφορά αυτή να μην κλείσει σήμερα, διότι στη Βουλγαρία δεν έχει λήξει το θέμα. Πολλό δε μάλλον που θεωρεί και αναφερόμενος ότι δεν πρέπει να κλείσει. Και το αναφέρει και στην επιστολή που μας έστειλε. Και αυτή η αναφορά νομίζω συνδέεται και με τις επόμενες δύο που θα εξετάσουμε λίγο αργότερα. Το θέμα δεν είναι μόνο η σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών, αλλά και κάτι στο πίσω δεν δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι η ε, ε, σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση παιδιών σε ιδρύματα. Αυτό δεν το προσέξαμε ίσως αρκετά και ε, εδώ πρόκειται για παιδιά με διανοητικές αναπηρίες που ακόμα είναι έγκλειστα σε ιδρύματα και ζουν σε πάρα πολύ εκτρές συνθήκε και συχνά δυστυχώς υφίστανται σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση. Και πιστεύω ε, ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της ε, ακριβώς το μηχανισμό παρακολούθησης και ελέγχου για να παρακολουθεί στενά όλες αυτές τις διαδικασίες που είναι τμήμα της καταπολέμησης του εγκλήματος και της μεταρρύθμισης της δικαιοσύνης. Η κυρία Ναντέλτσεβα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να συμφωνήσω και εγώ με την πρόταση που λέει να αφήσουμε ανοιχτή σήμερα την αναφορά αυτή, γιατί συνδέεται με άλλες τρεις σημαντικές πτυχές που συζητούμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα, πάρα πολύ ε, λεπτό και ευαίσθητο και φλέγον. Και θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε εμεί στο Κοινοβούλιο, στα κράτη-μέλη και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα και να βρούμε μία μόνιμη, μία βιώσιμη λύση. Θέλω να καλωσορίσω τη ε, λεγόμενη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Χρειάζεται εδώ μία ευρωπαϊκή στρατηγική με υψηλές προδιαγραφές και πρότυπα προστασίας των παιδιών, ειδικά τα παιδιά που ε, διαμένουν ε, σε ιδρύματα. Συμφωνώ με αυτά που είπε η κυρία Γιώτοβα. σε ιδρύματα ειδικέ αιστείες που φιλοξενούν παιδιά ε, και αν θέλετε να σας δώσω και πληροφορίες κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Και μια που μιλούμε και για το μηχανισμό ελέγχου και παρακολούθησης ε, για τη Βουλγαρία, ε, θέλω να πω ότι ε, φέτος για πρώτη φορά μετά την αλλαγή κυβέρνησης, η έκθεση του μηχανισμού παρακολούθησης και ελέγχου αναφέρει προόδους στη Βουλγαρία, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις δραστηριότητες των βουλγαρικών δικαστηρίων που εξετάζουν ε, περιπτώσεις στις οποίες ενέχονται υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενθαρρύνει τη χώρα να κάνει μεταρρυθμίσεις στον ποινικό κώδικα ε, και προχωρεί σε αλλαγές. Έχουν γίνει πολλά σημαντικά βήματα. Και ένα από αυτά ήταν η αύξηση των Από τριετή φυλάξη έγινε πενταετής. Και θα πρέπει να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στον τομέα αυτό με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει όμως να ασχοληθούμε περισσότερο με αυτό το θέμα και ε, να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στο πρόβλημα οι αρμόδιες αρχές για να επιταχυνθεί και η επίλυση του προβλήματος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους. Θέλετε το λόγο. Είναι προφανές ότι παραβιάζονται προκειμένου σε περιπτώσεις αυτές, δεν στέκω σε αυτή την περίπτωση μόνο, παραβιάζονται ανθρώπινα δικαιώματα και μάλιστα υπό επιβαρυντικές περιπτώσεις και υπό επιβαρυντικές περιστάσεις. Πρώτον, λόγω της ιδιότητος του δράστη, ο οποίος ε, καταχράτε τη δεσπόζουσα θέση της εποπτείας που έχει σε ανήλικα παιδιά και δεύτερον λόγω του γεγονότος ότι τα παιδιά αυτά έχουν πρόβλημα νοητικό. Συνεπώς θεωρώ ότι πρέπει να μείνει ανοιχτό το θέμα και όχι μόνο να μείνει ανοιχτό. Επειδή άκουσα ότι η υπόθεση δεν έχει κρυθεί τελεσίδικα, θα έλεγα να γίνει μια επιστολή στις δικαστικές αρχές της χώρας, στο ανώτατο δικαστήριο της χώρας αυτής, στο οποίο να τονίζουμε σαν Επιτροπή και σαν Ευρωκοινοβούλιο, σαν Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου, την ιδιαίτερη ευαισθησία μας που έχουμε πάνω στο θέμα και το γεγονός ότι παρακολουθούμε την περίπτωση. Εις τρόπον ώστε ε, να σκεφτούν πάρα πολύ καλά το τι θα κάνουν και οι δικαστές. Ξέρω πως σκέπτονται οι δικαστές, ιδιαίτερα σε βαλκανικές χώρες, και ξέρω πόσο ουσιαστική θα είναι η παρέμβασή μας εάν κάνουμε μια τέτοια παρέμβαση στο ε, ανώτατο δικαστήριο αυτής της χώρας. E Άλλοι τρει ζητούν το λόγο, αλλά σε 7 λεπτά έρχεται η Επίτροπο Ρέντινγκ. Παρακαλώ λοιπόν να είστε σύντομοι. Θα πρέπει δεν να διακόψουμε και τη συζήτηση των άλλων ε, αναφορών μεταξύ των οποίων έχουμε μία όπου ο υπογράφων είναι παρόν. Λοιπόν, παρακαλώ να είστε σύντομοι και να ολοκληρώνουμε αυτό το σημείο πριν έρθει ε, η Επίτροπος, κύριος Μπάιον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να σας χαιρετήσω μετά από ε, ε, ε, μια εξαιτή διακοπή πανακάμπτω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είναι η πρώτη συνεδρία στην οποία μπορώ να συμμετέχω ως αναπληρωτής. Έχω σπουδάσει νομική, έχω διατελέσει και δικηγόρος και με απασχολούν αυτά τα νομοθετικά ζητήματα και εργάζομαι σε αυτά. Θα παρακαλούσα να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά. Είμαι δε και στην Επιτροπή Πολιτισμού. Και η Επιτροπή Πολιτισμού ε, συζητά αυτό τον καιρό αυτή την απόφαση πλαίσιο, αλλά όχι μόνο η Επιτροπή Πολιτισμού και άλλα αρμόδια όργανα. Και η θέση του αναφερομένου ποια ήταν. Το πρόβλημα έχει να κάνει λιγότερο με τις ποινικέ κυρώσεις, αλλά περισσότερο με τις βουλγαρικές αρχές. Δηλαδή, ότι υπάρχει μια ανομία στη χώρα, δεν εφαρμόζονται οι νόμοι, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ε, πολιτικούς υψηλού βελνεκούς και υψηλόβαθμους αξιωματούχους της χώρας. Λοιπόν, παρακαλώ να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά και θα τα ξαναπούμε όταν θα έχουμε περισσότερα στοιχεία και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων επιτροπών. Ο συνάδελφος Γιάρ, παρακαλώ. Μια πρόταση μόνο συμπληρωματικά. Και εγώ θέλω να διατηρηθεί ανοιχτή η αναφορά, θα παρακαλούσα όμως να μην αναφερόμαστε μόνο στο δικαστήριο, αλλά να ε, ζητήσουμε να αποφανθεί, να γνωμοδοτήσει και η βουλγαρική κυβέρνηση. Θα παρακαλούσα να έχουμε και μια γνωμοδότηση της βουλγαρικής κυβέρνησης. Ωραία, αφήνουμε ανοιχτό το, το, το, ανοιχτή την αναφορά και μπορούμε να τη δούμε και αύριο στους συντονιστές. Επόμενη αναφορά. Λοιπόν, δίνω το λόγο στον υπογράφοντα. Κάρμεν Γκέρκα έχει το λόγο. Χαίρετε. Έχω ένα γιο που λέγεται Ρόμπερτ, είναι 14 ετών και έχει διαγνωστεί αυτιστικός. Το 2003 ίδρυσα μία ένωση, ένα σύλλογο με άλλους γονείς και ε, σήμερα έχει 50 μέλη και στο Γιάσο και σε ε, άλλες πόλεις είναι γονείς αυτιστικών παιδιών. Έχω κάνει πολλά στη χώρα μου για να ε, ευαισθητοποιήσω την κοινή γνώμη για τα άτομα με ε, αναπηρίες. Έχω κάνει πολλές αναφορές σε υπουργούς, σε κυβερνητικούς αξιωματούχους και όπου δει. Έχω κάνει και μια αναφορά πέρσι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουν λυθεί τα προβλήματά μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην απόφαση τη το έχει ξαναπεί και τονίσει ότι η Ρουμανία έχει υπογράψει πολλέ διεθνεί συμφάσεις, έχει ε, θεσπίσει και νόμου για τα άτομα με αναπηρίε. Θα ήθελα όμω να με καταλάβετε, ε, η νομοθεσία ε, Απλώ είναι ένα γενικό ευχολόγιο. Συγκεκριμένα δεν αναφέρεται τίποτα για την εφαρμογή. Τι γίνεται με του αυτιστικού, με ανθρώπου που έχουν νοητική αναπηρία, που είναι βαριά αναπηροί, δεν μπορούν να πάνε στο σχολείο τα παιδιά, δεν έχουν ειδική μεταχείριση, δεν έχουν ιατρική περίθαλψη, είναι πάυτοχες οι οικογένειές τους και δεν γίνεται και η διάγνωση σωστά. γιατί χρησιμοποιούν λαθασμένα κριτήρια για τη διάγνωση και δεν υπάρχουν και ειδικέ υπηρεσίε για τα παιδιά αυτά τα οποία ζουν απομονωμένα μέσα στι οικογένειέ του. Ενώ έχουν δικαιώματα τα οποία προβλέπουν και το Σύνταγμα και το άρθρο 14 της συνθήκης, μάλλον του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων που είναι όμως παράρτημα της συνθήκης. Τα παιδιά αυτά λοιπόν όχι μόνο δεν πηγαίνουν στο σχολείο ή δεν ε, ε, αντιμετωπίζονται από ειδικού γιατρούς αλλά δεν ενημερώνονται καν. Και από τότε που εγώ κατέθεσα την αναφορά, κατέβαλα προσπάθειε να αλλάξει η νομοθεσία στην ίδια μου τη χώρα για να διασφαλιστούν αυτά τα δικαιώματα των παιδιών με αναπηρίες. και έχω και υποστήριξη 100 με κυβερνητικών οργανώσεων στη χώρα μας. Αλλά εφιστάμεθα και διακρίσεις. Ο κόσμος δεν πληρώνεται, που είναι λιγότερο από 100 ευρώ ε, ο μισθός. Ε, για τους γονείς ομιλώ, ε, οι οποίοι γονείς αναγκάζονται τελικά να παραμένουν άνεργοι γιατί πρέπει να κάθονται σπίτι τους να φροντίζουν τα παιδιά τους που έχουν αναπηρίες. Και ε, κάτι άλλο που έρχεται να προσθεθεί επιβαρυντικό. Ε, υπάρχουν ιδρύματα μένα, αλλά πολύ λίγα, αλλά δεν ε, υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό ε, για να φροντίζει τα παιδιά αυτά και νοσηλευτικό και γενικότερο. Και η κατάσταση χειροτερεύει και μάλιστα σε επίπεδα χειρότερα της εποχής πριν το 89. Και σας είπα ότι ο μισθός είναι 100 ευρώ. Ε, εάν κάποιος ε, νοσηλευτής φροντίζει ε, δύο άτομα με αριά αναπηρία παίρνει 100 ευρώ. Εάν φροντίζει ένα μόνο, του κόβουν στα δύο το μισθό. Παίρνει μόνο 50 ευρώ. Και αυτά ο Δήμο. έτσι οι αρμόδιε αρχές της χώρα. Χρειάζεται λοιπόν μια νέα στρατηγική για την Ευρώπη, έτσι ώστε οι κοινωνικοί λειτουργοί, οι νοσηλευτέ να ε, ευαισθητοποιούνται για να καταλαβαίνουν και οι ειδικοί, το προσωπικό του ιατρικό, ε, ποια είναι η ανάγκη των παιδιών αυτών. Ε, στη Ρουμανία το κράτος δίνει το μισό του αντίστοιχου ευρωπαϊκού για τέτοιες υπηρεσίες πρόνοιας παρόλο που είναι η ε, πιο φτωχή χώρα ε, η Ρουμανία. Ο Ρόμπερτ, ο γιο μου λοιπόν που είναι 14χρονο, δεν μιλάει, αλλά μιλάω εγώ εξ ονόματό του και θέλω να μα βοηθήσετε. Και παρακαλώ την Επιτροπή ε, σας να μας υποστηρίξει πολιτικά. Δηλαδή στείλτε κάποιο γράμμα στις αρχές, στις αρμόδιες και στο Υπουργείο Απασχόλησης Κοινωνικών Υπηρεσιών κοινοποίηση στον Πρωθυπουργό. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ε, τα ε, παιδιά αυτά χρειάζονται φροντίδα. Οι εργαζόμενοι ε, που ασχολούνται και φροντίζουν τα παιδιά αυτά θα πρέπει να αναμείβονται και αξιοπρεπώς. Και επίσης κάτι άλλο που χρειάζεται είναι βελτίωση τη νομοθεσία, έτσι ώστε τα παιδιά αυτά να τη χάνουν τη σωστή φροντίδα, προστασία, να πηγαίνουν σχολείο, να ε, τους βλέπουν οι γιατροί. Έχουν το δικαίωμα τα παιδιά αυτά σε αυτή ε, την αντιμετώπιση. Και καλούνται να απαντήσουν λοιπόν οι ρουμανικές αρχές και θα παρακαλούσα και τους ε, ε, Ρουμάνους βουλευτές και τους άλλους ευρωβουλευτές να μας υποστηρίξουν. Συζητήστε το αυτό το θέμα, χρειάζεται λύση το συντομότερο. Σας παρακαλώ βοηθήστε μας για να βοηθήσουμε εμείς τα παιδιά μας να έχουν μια φυσιολογική ζωή. Γιατί στο κάτω-κάτω ευρωπαϊκή χώρα είναι και η Ρουμανία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ για την αναφορά σας. Όπως σας είχα πει, δεν θα ακολουθήσουμε πλέον την ημερήσια διάταξη. Θα ήθελα να χαιρετήσω την Επίτροπο Ρέντινγκ που έχει έρθει στην Επιτροπή μας, στην Επιτροπή Αναφορών. Θα ήθελα να της δώσω αμέσως λοιπόν το λόγο. Η Επίτροπος Ρέντινγκ αποδέχθηκε την πρόσκλησή μας να συμμετέχει στις εργασίες της Επιτροπής μας προκειμένου να αναφερθεί σε ζητήματα τα οποία εμείς σε καθημερινή βάση καλούμεθα να εξετάσουμε. Η Επίτροπος Ρέντινγκ ήδη πριν από μερικά χρόνια είχε ασχοληθεί πολύ άμεσα με τα ζητήματα αυτά και γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι σημαίνει να προεδρεύει κανείς σε μια τέτοια επιτροπή και τι σημαίνει να καταφέρει, να, να καταφέρει ουσιαστικά να καλύπτει όλα τα ζητήματα της ημερήσιας διάταξης. Πριν από 20 χρόνια, κυρία Πρόεδρε, πριν από 20 χρόνια προείδρευσα της Επιτροπής αυτής και πρέπει να σας πω ότι κατάφερα να μάθω πολλά για τα ευρωπαϊκά προβλήματα, για το ζήτημα της ηθαγένειας, για το τι μπορεί να κάνει κανείς για να επιλύσει τα προβλήματα αυτά. Κατά τη διάρκεια λοιπόν των τριών ετών που ασχολήθηκα με την Επιτροπή, κατάφερα πραγματικά να γνωρίσω καλύτερα τα προβλήματα αυτά που συναντούν οι πολίτες. Προβλήματα που ήταν κυρίως στην εποχή εκείνη διασυνοριακά, διασυνοριακής φύσης και προβλήματα τα οποία με τη μορφή αναφορών υποβάλλονταν στην Επιτροπή Αναφορών. Και εκείνη την εποχή τότε διοργανώθηκαν και οι πρώτες συναντήσεις μεταξύ του Επικεφαλής Επιτροπής Αναφορών και του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, ο οποίος μέχρι τότε δεν είχε έρθει σε επαφή με την Επιτροπή Αναφορών και δεν προβλεπόταν κάτι τέτοιο, αλλά τελικά έγινε και από τότε επισημοποιήθηκε αυτή η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ Επιτροπής Αναφορών και Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και ζήτησα κάτι τέτοιο γιατί συνειδητοποίησα ότι πάρα πολλές αναφορές που φτάνουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είχαν να κάνουν τόσο πολύ με το κοινοτικό δίκαιο όσο με την εθνική νομοθεσία. Και γι' αυτό το λόγο θεώρησα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτή η καλή σχέση εργασίας με τους εθνικούς συνηγόρους του πολίτη, στους οποίους θα μπορούσαμε να δίνουμε και άμεσα αναφορές που φτάνανε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου οι αναφορές αυτές να επιληθούν σε εθνικό επίπεδο, σε επίπεδο κράτους μέλους. Και θα θυμάμαι, θυμάμαι ότι κατά τη διάρκεια της εποχής εκείνης είχαμε και τη Μέρη Μπανότη, την πρώτη διαμεσολαβητή για την απαγωγή των παιδιών. Ήταν συναδελφός μου και χρειάστηκε να καταβάλει πολλές προσπάθειες προκειμένου να δημιουργηθεί η υπηρεσία αυτή. Δεν αναφέρομαι όμω πλέον στο παρελθόν, πολύ συχνά ξέρετε με τους ηλικιωμένου του κάνετε μια ερώτηση για το παρελθόν και αρχίζουν να διηγούνται ολόκληρη ιστορία. Προτιμώ να μιλήσω αυτή τη στιγμή για το μέλλον. Ξέρω κυρία Πρόεδρε ότι προβλέπετε στην ημερήσια διάταξη το ζήτημα της προστασίας των παιδιών, το διάφορα διασυνοριακά ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα δικαιώματα των παιδιών και το ζήτημα της ηθαγένειας. Υπάρχουν διάφορε προτάσει και μελλοντικέ προτάσει Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να χρησιμοποιείται μεγαλύτερη διαμεσολάβηση κάθε φορά που έχουμε οικογενειακέ διενέξει που έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα. Θα ήθελα να σα υπενθυμίσω ότι έχουμε ήδη μία οδηγία όσον αφορά την ε, διαμεσολάβηση, η οποία θα πρέπει να εφαρμοστεί τον Μάιο του 2011, θα πρέπει ουσιαστικά να μεταφερθεί στην Εθνική Νομοθεσία και βασίζομαι πολύ στην οδηγία αυτή γιατί πιστεύω ότι πάρα πολλές ε, υποθέσεις θα μπορούσαν να επιληθούν μέσω της ε, διαμεσολάβησης και ότι δεν χρειάζεται πλέον να προσφύγουμε αναγκαστικά στο δικαστήριο. Επίση, ε, βλέπω ότι ζητήσατε να διεξαχθεί μια μελέτη, μια μελέτη η οποία κάνει πολλές συστάσεις προκειμένου να αναπτυχθεί περισσότερο ο κανονισμός Βρυξέλλες 2α και προκειμένου να έχουμε κάποιες κοινέ ελάχιστες προδιαγραφές όσον αφορά την γονική ευθύνη. Ενδεχομένω να έχετε δει και το πρόγραμμα εργασία Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου προβλέπεται αναθεώρηση του κανονισμου βρυξελλες Βρυξέλλε 2α. Προβλέπεται αυτό για το 2013. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα είμαστε τότε στο τέλος της διαδικασίας. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να αναλύσουμε τι πηγαίνει καλά, τι λειτουργεί καλά στα πλαίσια του κανονισμού και τι θα χρειαστεί αργότερα να τροποποιηθεί. Είδα και τις συστάσεις λοιπόν της μελέτης που ζητήσατε και συμφωνώ ότι όντως θα πρέπει να φτάσουμε σε, κάποιους, σε κάποιες κοινέ ελάχιστες προδιαγραφές όσον αφορά την αναγνώριση και την εφαρμογή των αποφάσεων που έχουν να κάνουν με την γονική μέρημνα. Στόχος μου επίσης είναι να διακοπεί η διαδικασία να εξυμπήσει. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρχει μία κοινή εφαρμογή του κανονισμού αυτού που θα μπορούσε να οδηγήσει και σε μία μείωση των απαγωγών των παιδιών. Επίσης πρέπει να ασχοληθούμε με το ζήτημα των διεθνών διαζυγίων και προτιμάζουμε και έναν κανονισμό σχετικό. Αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε την διαδικασία της ενδυναμωμένης συνεργασίας. Έχουμε 14 κράτη-μέλη που θέλουν να εμπλακούν στη διαδικασία αυτή. Πολλές φορές και στις περιπτώσεις αυτές έχουμε άμεση προσφυγή στα δικαστήρια και τελικά είναι ο πιο ισχυρός, αν θέλετε, ο πιο ισχυρός διάδικος αυτός, ο οποίος καταφέρνει να κερδίσει την ε, κυδαιμονία του παιδιού. Εμείς θα θέλαμε να σταματήσει η διαδικασία αυτή και να έχουμε μια διαδικασία πολύ πιο ισορροπημένη, η οποία να μην ευνοεί τον έναν τον άλλον διάδικο, τον, ένα, τον άλλον γονέα συγκεκριμένα. Προτού προχωρήσουμε όμως σε μια αλλαγή των κανόνων, παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή πώς λειτουργεί ο κανονισμός Βρυξέλλες 2α στα κράτη-μέλη. Προσπαθούμε να εξετάσουμε συγκεκριμένα διάφορες ε, καταγγελίες που έχουν κάνει οι ίδιοι Ευρωπαίοι πολίτες Ξέρετε ότι τα παράπονα αυτά, οι καταγγελίες αυτές μπορούν να οδηγήσουν ακόμα και στη διαδικασία επιπαραβάση εναντίον ενός κράτους μέλους. Αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ένα κράτος μέλος δεν τα αποκρίνεται στις υποχρεώσεις του στα πλαίσια της συνθήκης. Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η διαδικασία επιπαραβάση αποτελεί έναν από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για τη διόρθωση της μη καλής εφαρμογής ενός κανονισμού. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για την κακή εφαρμογή κανονισμού και όχι για την ε, ερμηνεία του κανονισμού από το ένα ή το άλλο δικαστήριο. Αναφέρομαι συγκεκριμένα στην περίπτωση που ένα κράτος μέλος δεν εφαρμόζει σωστά τον κανονισμό. Στην περίπτωση αυτή, όπως σας εξήγησα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να προσφύγει κατά κράτους μέλους στο δικαστήριο. Μέσω λοιπόν της έντονης αυτής επιτήρησης και παρακολούθησης προσπαθούμε να δούμε πώς εφαρμόζεται ο κανονισμός στα κράτη-μέλη και συγκεκριμένη Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εντοπίσει ένα στοιχείο το οποίο θα μπορούσε να αρχίσει να εφαρμόζεται χωρίς να χρειάζεται να προχωρήσουμε σε μια αναθεώρηση της νομοθεσίας. Και αναφέρομαι αυτή τη στιγμή στην ε, κατάρτιση, στην εκπαίδευση των εμπειρογνωμόνων. Πρέπει ουσιαστικά να έχουμε περισσότερου εμπειρογνώμονε στα κράτη-μέλη, νομομαθεί, που να είναι σε θέση να καταλάβουν καλύτερα τι διασυνοριακέ υποθέσει. Χρειαζόμαστε δικαστέ, νομικού, δικηγόρου, οι οποίοι να είναι σε θέση να καταλάβουν και να εξετάσουν καλά τι περιπτώσει αυτέ. Ξέρετε ότι έχουμε, όπως σας είπα, τον κανονισμό Βρυξέλλες 2α, ο οποίος αρχίζει και εφαρμόζεται στα κράτη-μέλη, θα επενδύσουμε περισσότερο, αν θέλετε, στην κατάρτιση των νομομαθών, προκειμένου να σε θέση να εφαρμόσουν καλύτερα τον κανονισμό αυτό. Δεύτερο τώρα ζήτημα, δικαιώματα των παιδιών. Θα θυμάστε ότι κατά τη διάρκεια της ακρόασης που διοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το ζήτημα αυτό ετέθη και σας είχα αποσχεθεί τότε ότι θα αποτελούσε προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με συγκεκριμένα μέτρα όσον αφορά την προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών. Τα μέτρα αυτά για τα δικαιώματα των παιδιών δεν μπορούν να αποτελέσουν αρμοδιότητα ενός μόνο επιτρόπου, αλλά πρέπει να αποτελέσουν ε, οριζόντιο μέλημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα πρέπει να εισαχθούν σε όλες τις δράσεις και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης βάσει του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων την περίοδο αυτή δεν θα έλεγα ότι προετοιμάζω μια ανακοίνωση. Έχω ουσιαστικά ολοκληρώσει μια ανακοίνωση η οποία θα δημοσιευθεί τις επόμενες εβδομάδες και θα αποτελεί ουσιαστικά το πρόγραμμα δράσης για το πώς θα εργαστούμε για την προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Κυρίως ε, σε σχέση με τον ε, τομέα της δικαιοσύνης όπου θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε ένα δικαστικό σύστημα φιλικό προς τα παιδιά. Θέλουμε να ενισχύσουμε την προάσπιση των παιδιών στα πλαίσια των δικαστικών διαδικασιών και να ενδυναμώσουμε και το ζήτημα της ε, γονικής ευθύνης. Με ιδιαίτερη χαρά λοιπόν θα ήθελα να συζητήσω το ζήτημα αυτό με τους Ευρωβουλευτές από τη στιγμή βέβαια που θα είναι πλέον έτοιμη η ανακοίνωση αυτή και θα έχει υποβληθεί επίσημα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ακολουθεί η συνήθις κοινοβουλευτική διαδικασία και για την ανακοίνωση αυτή. Όσον αφορά την πληροφόρηση προς τους πολίτες και την επίλυση των προβλημάτων των πολιτών, σε συνεργασία με την κυρία Βάλεαν, τη συναδελφό σας, σήμερα το απόγευμα πήγα στην ετήσια Γενική Συνέλευση του δικτύου Europe Direct, Europe Direct Network. Το δίκτυο αυτό σε τήσια βάση λαμβάνει περίπου ένα εκατομμύριο αιτήματα για προβλήματα παντός είδους. Και έχουμε δημιουργήσει, αν θέλετε, μία κοινή πύλη, μία ενιαία θηρίδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της οποίας οι, Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να υποβάλουν τα αιτήματά τους, τα οποία στη συνέχεια διανέμονται σε όλα τα αρμόδια θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία καλούνται στη συνέχεια να απαντήσουν. Οι διασυνοριακές υποθέσεις αποτελούν περίπου 25.000 ετησίως. 25.000 ε, αιτήματα έχουν να κάνουν με διασυνοριακές υποθέσεις. Αιτήματα τα οποία φτάνουν ε, στο Europe Direct Network. Νομίζω ότι ε, οι αναφορές που φτάνουν σε εσά είναι περίπου 2.000 ετησίως. Καταλαβαίνετε λοιπόν ποιο είναι αν θέλετε το μέγεθος του προβλήματος το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Γιατί δεν υποβάλλουν όλοι αναφορές στην δική σας επιτροπή, ούτε στέλνουν όλοι αιτήματα στο Europe Direct. Επομένως, ε, αναφερόμαστε σε 27.000, καταλαβαίνετε ποιος μπορεί να είναι ο πραγματικός αριθμός αν να συμψηφίσουμε όλα αυτά τα αιτήματα και τις αναφορές. Και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο πρόεδρος Μπαρόσο, αποφάσισε ότι θα πρέπει να δοθούν πολύ συγκεκριμένε αποφάσεις στα προβλήματα αυτά. Δεν αρκεί αυτή τη στιγμή να βγάζουμε κάποιους θεωρητικούς λόγους, θα πρέπει να προχωρήσουμε σε συγκεκριμένα μέτρα. Και έχουμε επίση και την έκθεση του κυρίου Αλάν Λαμασούρα, έκθεση που υπέβαλε το 2008, στο οποίο καταγράφονται όλα τα εμπόδια τα οποία συναντούν οι πολίτες και δίνονται και πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα. Εμπόδια λοιπόν τα οποία συναντούν οι πολίτες κάθε φορά που θέλουν να ασκήσουν το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας. Και για αυτό το λόγο αυτή την εβδομάδα την Τετάρτη θα έχουμε μία ξεχωριστή διοργάνωση, ένα ειδικό γεγονός. Ξέρετε ότι θέλουμε να δυναμώσουμε περισσότερο την εσωτερική αγορά για οικονομικούς λόγους και κατά αυτόν τον τρόπο μόνο μπορούμε να ενισχύσουμε τη θέση μας σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να προωθήσουμε τις δικές μας επιχειρήσεις μέσω μιας πιο ενισχυμένης αγοράς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να γίνει κάτι τέτοιο, να διευκολυνθούν οι διασυνοριακές οικονομικές σχέσεις και γι' αυτό τον λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Τετάρτη θα υποβάλει εκ νέου νέες προτάσεις για την εσωτερική αγορά. Ο Επίτροπος Μπαρνιέ θα δώσει μια συνέντευξη τύπου, αλλά θα το συνοδεύει και ένας άλλος Επίτροπος, εγώ ίδια ουσιαστικά. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε ότι η εσωτερική αγορά δεν έχει να κάνει μόνο με επιχειρήσεις και με οικονομικά, έχει να κάνει και με τους ίδιους τους ανθρώπους στα πλαίσια της εσωτερικής αγοράς. Θα έχουμε λοιπόν και τις δύο πλευρές του ζητήματος αυτού να παρουσιάζονται ταυτοχρόνως τόσο την οικονομική πτυχή όσο και την πτυχή εκείνη που έχει να κάνει με την ηθαγένεια, με τους πολίτες. Πώς μπορούμε ουσιαστικά να καταρρύψουμε τα εμπόδια αυτά που υπάρχουν ένα προς ένα με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Θα αναφερθούμε σε 25 συγκεκριμένες δράσεις με συγκεκριμένες προθεσμίες. Δεν θα μιλάμε λοιπόν μόνο για θεωρητικές δεσμεύσεις μελλοντικέ, θα δίνουμε και ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα που θα προβλέπει συγκεκριμένε προθεσμίες για κάθε μία από τις 25 δράσεις στις οποίες αναφερθούμε. Θα δείτε δηλαδή πώς μέσα από συγκεκριμένες δράσεις θα καταρριφθούν ένα προς ένα όλα τα εμπόδια τα οποία συναντούν οι Ευρωπαίοι πολίτες κάθε φορά που θέλουν να προχωρήσουν σε μια ε, διασυνοριακή δράση, αν θέλετε, κάθε φορά που επιθυμούν ως φοιτητές, ως μαθητές, ως επιχειρηματίες να ασκήσουν τα δικαιώματά τους σε μια άλλη χώρα. Θα ήθελα επίσης να προτείνω το έτος 2013 ως ευρωπαϊκό έτος για τους Ευρωπαίους πολίτες. Ελπίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα υποστηρίξει την πρότασή μου αυτή. Μη μου πείτε αυτή τη στιγμή ότι απλώς προτείνω ένα ακόμα ευρωπαϊκό έτος. Κάνω την πρόταση αυτή γιατί πιστεύω ότι χρειαζόμαστε ένα τέτοιο ευρωπαϊκό έτος προκειμένου να καταφέρουμε να συντονίσουμε όλες αυτές τις δράσεις που θα πρέπει να λάβουν χώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε εθνικό επίπεδο γιατί δεν είναι δυνατόν να επιβάλλουμε μόνο από τις Βρυξέλλες τα δικαιώματα των πολιτών. Θα πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ του κοινοτικού και του εθνικού επίπεδου, αλλά και του τοπικού και του περιφερειακού επίπεδου. Αυτή λοιπόν θα είναι η στόχη του Ευρωπαϊκού Έτους για τους Ευρωπαίους πολίτες και ελπίζω ότι μπορώ να βασίζομαι στη δική σας υποστήριξη, στην υποστήριξη Επιτροπής Συναφορών. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας αυτή, σας ευχαριστούμε πολύ για όλες αυτές τις προτάσεις που εκφράσατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη αυτή τη σημαντικότητα εργασία που έχετε ήδη ξεκινήσει. Μπορεί τώρα να ξεκινήσει η συζήτηση με τους συναδέλφους. Ο κύριος Μποσινάρου πρώτος θέλει το λόγο, έτσι δεν είναι. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Χαίρομαι πάρα πολύ και με ενθαρρύνει ε, η τοποθέτησή σας. Αλλά νομίζω το πιο ε, ευνοϊκό που άκουσαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, πρόσφατα και το πιο εθελοντικό ήταν αυτό που είπατε το φτάνει πια. Η is enough. Και όντω η Ευρώπη μπορεί να έχει αποτελέσματα. Και σε ό,τι αφορά την Επιτροπή μας εδώ αναφορών, γνωρίζετε πολύ καλά την Επιτροπή αυτή και γνωρίζετε ότι τρία είναι τα στοιχεία ε, βάσει των οποίων είμαστε σε ε, διαρκή επαφή με τους πολίτες, αλλά προσπαθούμε να τους δώσουμε και απαντήσεις. Περιβάλλον, βιοπικιλότητα και ρήπανση, που είναι κατεξοχήν διασυνοριακά θέματα. Και θα ήθελα, σας παρακαλώ, να μας υποστηρίξετε κι εσείς. Σας παρακαλώ να δώσετε στην Ένωσή μας τα νομικά εκείνα εργαλεία που χρειάζεται για να αντιμετωπίζει σε διασυνοριακό επίπεδο ε, τα προβλήματα που σας ανέφερα προηγουμένως. Αυτό ήταν το πρώτο. Δεύτερον, χαίρομαι πάρα πολύ για τις τάσεις σας, για τις θέσεις που παίρνετε. όλο και περισσότερο ε, κερδίζουν έδαφος ε, πρόσφατα οι φωνές που ζητούν ε, λύσεις σε εθνικό επίπεδο. Γι' αυτό είναι και πιο σημαντικό εμείς οι Ευρωπαίοι, εμείς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εμείς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δίδουμε ευρωπαϊκές λύσεις για ευρωπαϊκά προβλήματα τα οποία αφορούν την καθημερινότητα των Ευρωπαίων πολιτών. Και θα ήθελα να αφαιρθώ σε κάτι το οποίο είναι όντως πάρα πολύ σημαντικό γίνεται μία απόπειρα είτε να περιορίζεται ε, είτε να ελέγχεται πολιτικά η ελευθεροτυπία, του, η ελευθεροτυπία σε κάποιες χώρες. Και εδώ αναφέρομαι ειδικά στη δική μου χώρα, τη Ρουμανία, όπου η ελευθερία του τύπου, κυρία Επίτροπε, θεωρείται ότι ε, πλήττει την εθνική ασφάλεια, λέει. Όταν είναι ο τύπος ελεύθερος, αυτό είναι εις βάρος εθνικής ασφάλειας. Τι στρατηγική είναι αυτή. Δεν θα δείτε ποτέ ε, κανένα ε, τέτοιο προηγούμενο. Συγγνώμη που κάνω τέτοια σκληρή αναφορά. Είναι αυτά πράγματα να λέγονται ότι η ελευθερία του τύπου βλάπτει την εθνική ασφάλεια της χώρας. Επίσης χαίρομαι πάρα πολύ για αυτά που είπατε για μια ειλικρινή σχέση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ευρω... Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να μπορέσουμε να οικοδομήσουμε και να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Φτάνουν τα λόγια. Έργα τώρα χρειαζόμαστε. Και είμαι βέβαιο ότι από κοινού θα μπορέσουμε να αποδώσουμε. Ευχαριστώ. Η ε, κυρία Γκρινή. Ευχαριστώ πολύ που δεχθήκατε κυρία Επίτροπε αυτή την πρόσκλησή μας. Πάντα χαίρομαι να συναντώ επιτρόπους. Πρόκειται για ένα ζήτημα για το οποίο έχετε μιλήσει πολύ για τα δικαιώματα των παιδιών εμείς πάντα πρέπει να βοηθάμε τον πιο αδύναμο, τον πιο μικρό και να επιλύνουμε τα προβλήματα του. Το πρόβλημα των παιδιών είναι από τα πιο, της προστασίας των παιδιών είναι από τα πιο παλιά που αντιμετωπίζουμε αλλά δεν βλέπουμε λύσεις. Πώς σκοπεύετε εσείς να τα προστατεύσετε για την εργασία ας πούμε από τις σεξουαλικές καταχρήσεις ε, τα ανάπηρα παιδιά, ε, η εκπαίδευση παιδεία για όλους να ενσωματωθούν στην αγορά εργασίας και στη στρατηγική 2020 για τη μείωση της φτώχειας. Όλες, αυτά, όλες αυτές οι πολιτικές βρίσκονται στη βάση των προβλημάτων των παιδιών. Εσείς μιλήσατε για το στόχο της διαμεσολάβησης, μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον αυτό. Μπορείτε όμως να βρείτε δεσμε, νομικώς δεσμευτικά μέτρα γιατί τα θέματα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά αλλά και λεπτά θέματα όταν βλέπουμε εμεί τα δικαίωμα επίσκεψη, το δικαίωμα στην επιμέλεια. Όλα αυτά τα θέματα είναι δύσκολα, υπάρχουν πάντοτε προβλήματα και τις ίδιες δυσκολίες αντιμετωπίζουν και οι δικαστές. Πολλές φορές η Επιτροπή μας των Αναφορών είναι άοπλη, διότι όλοι επικαλούνται την αρχή της επικουρικότητας, ε, όπου αρμόδια είναι τα κράτη-μέλη και εμείς δεν έχουμε δεσμευτικά μέτρα που να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε. Κύριο Σαμάνσκι. Άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή την τοποθέτησή σας και διάβασα και με ιδιαίτερη προσοχή την ανακοίνωση που μας στείλατε σήμερα για την αναφορά της κυρίας Κολόμπο. Γνωρίζω πολύ καλά αυτήν την αναφορά γιατί εξέτασα αντίστοιχες ε, αναφορές και στην προηγούμενη θητεία που αφορούσαν σε Πολωνούς πολίτες. Εκπλήσωμαι γιατί θεωρώ ότι η Κομισιόν αντιμετωπίζει τα πράγματα με ιδιαίτερη παθητικότητα. Σίγουρα εμείς ε, πρέπει να προασπίσουμε το θέμα των ε, δικαιοδοσιών σε εθνικό επίπεδο. Αλλά ας πούμε βλέπετε με τις δράσεις του Jugendamt όπου έχουμε διακρίσεις ε, Ευρωπαίοι πολίτες πρέπει λοιπόν εμείς να ή τουλάχιστον να, να προβληματιστούμε για το κατά πόσο αυτές οι δράσεις οδηγούν σε διακρίσεις. το Jugendamt λέει ότι το καλό και συμφέρον για το παιδί είναι να μάθει γερμανικά, να έχει στενή επαφή με το γερμανό γονιό. Αυτό όμως το μέτρο δεν οδηγεί σε μία διάκριση ε, υπέρ των Γερμανών και κατά των υπολείπων ο κανονισμός Βρυξέλλες 2α έχει, την, έχει στόχο ε, να βοηθήσει τους γονείς που χωρίζουν και που έχουν διαφορετική υπηκότητα μεταξύ τους. Όταν λοιπόν βλέπουμε εμείς το Jugendamt να οδηγεί, ε, να δημιουργεί μια δυσκολία σχέσεων ε, και πάντοτε υπέρ του Γερμανού γονιού ε, δεν υπάρχει ένα πρόβλημα. Πίστευω ότι η Κομισιόν κρατάει μια παθητική στάση και σε άλλες αναφορές ε, νύπτει τα σχήρα πάρα πολύ εύκολα. Πάντα μας θυμίζουν, ορίστε υπάρχουν οι εθνικές αρμοδιότητες, αλλά αυτές, αυτού του είδους οι καταστάσεις είναι καταστάσεις πολύ ε, πο, πο, πολύ σπάνιες και μόνο σε αυτές τις ε, περιπτώσεις ε, γίνεται τόσο έντονη αναφορά στην επικουρικότητα. Η κυρία Νεντέλτσεβα, εγώ δεν θέλω να περιορίσω την συζήτηση, αλλά αν αυτοπιθαρχηθούμε λίγο θα μπορέσει να μας απαντήσει η Επίτροπος. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, επιτρέψτε μου καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ σήμερα ενώπιόν μας και επιτρέψτε μου να εκφράσω και την ικανοποίηση και ε, τη χαρά μου για τη διαρκή μόνιμη επαφή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που καλλιεργείται και το επίπεδό της. Και Χαίρομαι για αυτό που είπατε ότι προτείνεται το 2013 να είναι το Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών και αξίζει να υποστηριχθεί αυτή η προσπάθειά σας από όλο το Κοινοβούλιο. Έχω δύο ερωτήσεις σήμερα, σύντομες. Ε, πρώτη ερώτηση. Λαμβάνουμε εδώ διάφορες αναφορές στην Επιτροπή μας σχετικά με α, παιδιά με αναπηρίες και τον αποκλεισμό που υφίστανται σε διάφορα κράτη-μέλη γνωρίζω και καταλαβαίνουμε ότι είναι καταπάτηση και άρνηση των βασικότερων θεμελιωδέστερων δικαιωμάτων τους αυτό. Και το γνωρίζετε. Ε, στα περισσότερα κράτη-μέλη διαπιστώνουμε ότι χρειάζονται επιπλέον μέτρα πέρα από την κοινωνική πολιτική. Εσείς έχετε συζητήσει, προτίθεστε να αναλάβετε κοινέ δράσεις με τον Επίτροπο Άντορ σε αυτό το τομέα, γιατί νομίζω ότι χρειάζεται μεγαλύτερη συνοχή και συνεργασία μεταξύ των δύο επιτρόπων και γενικότερα. Δεύτερη ερώτηση. Συζητούμε όλοι για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών σε περίπτωση που χωρίζουν οι γονεί του ε, και είναι από διαφορετικέ χώρε. Εγώ θα ήθελα να σα επιστήσω την προσοχή σε πάρα πολλέ ε, περιπτώσει διεθνών υιοθεσιών. Στην Ευρώπη πολλέ φορέ είναι πάρα πολύ μακροχρόνιε οι διαδικασίε και πάρα πολύ οδυνηρέ. Θα προτείνετε τίποτα ε, αν μη τι άλλο για τα διάφορα αρμόδια όργανα και για τις προθεσμίες που έτσι και αλλιώς ε, αυτά γράφονται στα επίσημα έγγραφα. Αλλά θα ήθελα να γνωρίσω τι προτάσεις έχετε για αυτό το θέμα των διεθνών υιοθεσιών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία ουκέν Ευχαριστώ πολύ κυρία Επίτροπε. Θα ήθελα να πω και εγώ ότι χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπουμε ενωπιών μας. Σας ευχαριστώ και για τα όσα μας είπατε. Παίρνω το λόγο για να υποστηρίξω τον συνάδελφο Μποστινάρου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πλέον και κρίσιμο τα βασικά θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, όπως περιγράφονται στη συνθήκη, την ίδια στη συνθήκη λέω, θα πρέπει να θεωρούνται τμήμα ενός δικαίου ε, που διέπει όλες τις χώρες επανειλημμένα βλέπουμε στην Επιτροπή μας, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσπαθεί να ξεφορτώνεται, για να το πω έτσι, ευαίσθητα θέματα. Τα παραπέμπει στην ε, επικουρικότητα. Και χαίρομαι για αυτά που λέτε πολύ έντονα για την καταπολέμηση των διακρίσεων των Ρωμά. Χαίρομαι που τα είπατε και που σας άκουσα. Στο μεταξύ έχει ίσως ξεχαστεί το θέμα και χαίρομαι και για αυτά που είπατε εδώ στο Κοινοβούλιο. Ήταν πάρα πολύ αποτελεσματικά και όσοι διαβάζουν ανάμεσα από τις γραμμές και σκέφτονται κατάλαβαν περί τίνος πρόκειται. Σας ευχαριστώ πολύ. Ξέρουμε ότι οι διακρίσεις είναι ένα θέμα πάρα πολύ βαρύ, έτσι σοβαρό που θα πρέπει να το συζητάμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να το αντιμετωπίσουμε. Και για την ελευθεροτυπία. Ακούω τι γίνεται στη Ρουμανία και έχω την εντύπωση ότι, ξέρω εγώ, αναστήθηκε ο Τσαουσέσκου. Τι γίνεται εκεί και έχει επαναφέρει το παλιό καθεστώς, το έχει αναστηλώσει, γιατί ε, γίνονται τρομακτικά πράγματα και ακούμε τρομερές ιστορίε. Και αν αυτό δεν είναι θέμα που απασχολεί όλα τα κράτη-μέλη, τι να πούμε. Δεν λέω ότι θέλουν να φημώσουν τον τύπο, αλλά τον περιορίζουν πάρα πολύ τον ελεύθερο τύπο. Λοιπόν, είναι θέμα που μας αφορά όλους. Και διακυβεύεται και η δική μας αξιοπιστία. Σας ευχαριστώ και ε, κάποια στιγμή να έρθει αυτό το θέμα και στη δική μας ατζέντα. Και όχι να αφήνουμε την ευθεροτυπία στην Ιταλία, στη Ρουμανία. Κάποια μέρα μπορούμε να τη βρούμε μπροστά μας όλοι μας. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπουσουτήλ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να καλωσορίσω την κυρία Επίτροπο ενώπιον μας και να την ευχαριστήσω για την παρουσία της και την παρουσίασή της. Συμφωνώ και εγώ και την υποστηρίζω για την πρόταση το 2013 <coughs> να κηρυχθεί έτος των Ευρωπαίων πολιτών. Νομίζω ότι θα δώσει αυτό μια πολύ σπουδαία όθηση ε, στα δικαιώματα των πολιτών και θα ενδιαφερθούν περισσότερο οι πολίτες να μάθουν ποια είναι τα δικαιώματά τους. Ε, για τις καταγγελίες των πολιτών ε, διαμαρτύρονται οι πολίτες ότι είναι πολύ μεγάλες οι προθεσμίες. Ας πούμε, όταν ένας πολίτης καταγγέλει κάτι ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη δική μας Επιτροπή, περνάει πάρα πολύ καιρό μέχρι να δοθεί συνέχεια. Γνωρίζω, κυρία Αντιπρόεδρε, ότι ε, σας ενδιαφέρουν πολύ τα δικαιώματα των πολιτών, αλλά τι προτίθεστε να κάνετε ώστε να μειωθούν αυτοί οι ε, χρόνοι, οι τρομερέ καθυστερήσει. Δηλαδή, ο χρόνο που περνάει από τη στιγμή που κάνει την καταγγελία του ένα πολίτη μέχρι να απαντηθεί, περνάει πάρα πολύ ε, Για το θέμα το Ρωμά στη Γαλλία, δράσατε πάρα πολύ γρήγορα. Και καλώ ε, πράξατε. Ε, συγχαίρω, αλλά δεν θα πρέπει ε, αυτό να ισχύει και για όλου του πολίτε. Ένα δεύτερο που έχω να θέσω. Για τον νόμο για τα δικαιώματα των παιδιών, όπως είπε η συνάδελφος ε, Γκρουνή. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία για τους ανήλικες είναι πάρα πολύ κατακαιρματισμένη. Έχουμε κοινωνική νομοθεσία, ε, ε, εργατική νομοθεσία και ένα νέο νόμο που προσπαθούμε τώρα να περάσουμε για τη σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών. Δεν υπάρχει όμως ένας ενιαίος ευρωπαϊκός νόμος που να καλύπτει όλο το φάσμα των δικαιωμάτων των παιδιών. Νομίζω λοιπόν ότι κάτι τέτοιο θα ήταν πολύ σημαντικό και σας παρακαλώ να το σκεφτείτε και αυτό. Ε, μέχρι το τέλος της θητείας σας να έχετε αφήσει ε, πίσω ε, μια πολύ σημαντική κληρονομιά για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα δικαιώματα των παιδιών. Τέσσερις έχουν ζητήσει ακόμη το λόγο και μας λείπουν 14 λεπτά για να τελειώνουμε με την, και με την απάντηση της Επιτρόπου. Σύντομη λοιπόν. Κύριος Μπάιενς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ναι, θα είμαι σύντομος. Συμφωνώ και εγώ με τους προλαλήσαντες. Θέλω να καλωσορίσω και να συγχαρώ και την Επίτροπο. Θα σας υποστηρίξουμε και εγώ και ολόκληρη η Ουγγρική Αντιπροσωπεία στην προσπάθεια αυτή να ε, κηρυχθεί το 2013 το έτος του Ευρωπαίου Πολίτη. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Τι στόχους έχετε στα πλαίσια της καταπολέμησης της παιδικής πορνογραφίας και της καταπολέμησης σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών. Και μια άλλη ερώτηση έτσι πιο προσωπική θα ήθελα να σας κάνω. Επί μια τετραετία ε, διατέλεσα επικεφαλής μιας επιτροπής στην Ουγγαρία όπου είχαμε πάρα πολλά προβλήματα, έτσι σε ένα επαρχιακό επίπεδο. Είχαμε προβλήματα γιατί δεν υπήρχε ευρωπαϊκή στρατηγική για τα παιδιά με αναπηρία. Και ε, εξ όσων γνωρίζω, έχετε και ε, άλλες προτάσεις για την ευρωπαϊκή στρατηγική για παιδιά με αναπηρίες. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπέλντερ. Μπέλντερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν ζήτησα το λόγο. Η κυρία Χέρκο ε, ήθελε μάλλον το λόγο. Εγώ δεν ζήτησα το λόγο. Λοιπόν, δύο τοποθετήσεις. Βάλιαν. Σύντομα, Επίτροπε, συγχαρητήρια. έχετε την υποστήριξή μου και όλη τη πολιτική ομάδα. Το χαρτοφυλάκιο σα είναι πολύ κρίσιμο. Και έχω την εξερώτηση. Λαμβάνοντα υπόψη και το προηγούμενο χαρτοφυλάκιο που είχατε και την τωρινή σα θέση. Ε, πώς συνδυάζονται αυτά τα δύο χαρτοφυλάκια. Ε, κυρία Γιώτοβα, ε, ορίσατε κύριε Επίτροπε. Εμείς οι σοσιαλιστές εγκρίναμε ε, το διορισμό σας σε αυτό το χαρτοφυλάκιο, γιατί θέλαμε πραγματικά έναν επίτροπο που να ασχολείται με ανθρώπινα δικαιώματα και ιδίως με τα δικαιώματα των ανηλίκων. Σήμερα συζητήσαμε ε, στην Επιτροπή μας ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό ε, και κρίσιμο που έχει να κάνει με ανάπηρα παιδιά. Εξ όσων γνωρίζω, είναι ένα θέμα που σας ενδιαφέρει και εσάς τα δικαιώματα των παιδιών και προετοιμάζεται ειδική ανακοίνωση σχετικά. Θα ήθελα όμως να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στα παιδιά με αναπηρίες. Δεν έχει έρθει η ώρα να βεβαιωθούμε ότι και τα δικά τους δικαιώματα γίνονται σεβαστά. Να γίνεται μια ειδική και συγκεκριμένη αναφορά και σε αυτά. Γιατί σήμερα μιλήσαμε για ιδρύματα όπου φιλοξενούνται παιδιά με αναπηρίες και σε ορισμένε χώρες είναι πολύ δύσκολε οι συνθήκε και της διαβίωσης των παιδιών αλλά και τη εργασία του προσωπικού που απασχολείται εκεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δίνω το λόγο τώρα στην Επίτροπο Ρέντινγκ. Την ευχαριστώ πολύ. Και ελπίζω σε λίγα λεπτά να μπορέσει να απαντήσει στις ε, τόσες ε, πολλές ερωτήσεις που της ετέθησαν. Ε, μα είναι αδύνατη αυτή η αποστολή. Θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι μπορώ, όσο πιο σύντομα γίνεται, γιατί υπάρχουν ορισμένοι βουλευτές που έχουν θέσει πάνω κάτω τις ίδιες ερωτήσεις. Κατάλαβα ότι α, πολλοί πιστεύετε ότι το 2013 πρέπει να ανακηρυχθεί έτος των Ευρωπαίων πολιτών. Επομένως θα συνεργαστούμε για να αποτελέσει το έτος αυτό ένα πολύ αποτελεσματικό έτος γιατί εσείς είστε η πραγματικά πιο αποτελεσματική εταίροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εσείς γνωρίζετε τους πολίτες. Οι πολίτες προέρχονται από τη δική σας εκλογική περιφέρεια. Είναι πολύ σημαντικό ουσιαστικά να τους βοηθήσετε να εισακουστούν στις Βρυξέλλες. Από την εμπειρία μου ως πρόεδρος της Επιτροπής αυτής γνωρίζω πόσο σημαντικό είναι το ζήτημα που έχει να κάνει με το περιβάλλον. Πριν από 20 χρόνια μιλούσαμε κυρίως για την κατασκευή δρόμων και αναφερόμασταν ε, στο πρόγραμμα Natura για την προστασία του περιβάλλοντος. Τώρα μιλάμε κυρίως για την βιοπικιλότητα και για τη μόλυνση. Είναι ξεκάθαρο τα φαινόμενα αυτά έχουν διασυνοριακές επιπτώσεις και ο συνάδελφος που είναι υπεύθυνο για το ζήτημα του περιβάλλοντος, καθώς επίσης και ο συνάδελφος που είναι υπεύθυνο ε, για το ζήτημα της ενέργειας και οι δύο ασχολούνται με τα διασυνοριακά αυτά ζητήματα. Και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας όταν λέτε ότι χρειαζόμαστε ευρωπαϊκές λύσεις κατά των εθνικιστικών τάσεων. Οι τάσεις αυτές είναι ουσιαστικά πολύ κοντόφθαλμες. Αν δείτε τι γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο, τότε συνειδητοποιείτε ότι και κάποια μεγάλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ουσιαστικά μικρά. Να μην αναφερθούμε και στα μικρά βέβαια. Και γι' αυτό το λόγο αποφασίσαμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανακινήσουμε την πολιτική εσωτερικής αγοράς για τις επιχειρήσεις τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις και βέβαια να προωθήσουμε μέσω της πρότασης αυτής και τους πολίτες. Θέσατε επίσης ένα πολύ συγκεκριμένο ερώτημα όσον αφορά την ε, ελευθεροτυπία, την ελευθερία των ε, μέσων ενημέρωσης. Είμαι ανήσυχη. Ανήσυχη για τα όσα συμβαίνουν στα κράτη-μέλη στα οποία αναφερθήκατε εν γέννη, καθώς επίσης και σε κάποια άλλα κράτη-μέλη πιο συγκεκριμένα. και σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω με αυτό το οποίο αναφερθήκατε εσείς, αυτό που λέει η κυβέρνησή σας. Τα ελεύθερα μέσα ενημέρωση είναι εγγύηση της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Ορισμένα, ορισμένα μέσα ενημέρωση μπορεί να υπερβάλλουν, αλλά έχουμε νόμους οι οποίοι θα πρέπει να προστατεύουν τα μέσα ενημέρωση, αλλά και τα δικαιώματα των πολιτών σε σχέση με τα μέσα ενημέρωση. Το να λέμε όμως ότι τα ελεύθερα μέσα ενημέρωση μπορούν να αποτελέσουν αδύναμο σημείο της εθνικής ασφάλειας, αυτό θα έπρεπε να αποδειχτεί στην πράξη για να αναλυθεί και νομίζω ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να αποδειχτεί. Ήμουνα επίτροπο υπεύθυνη για τα μέσα ενημέρωση για 10 χρόνια και θεωρώ ότι τα ελεύθερα μέσα ενημέρωση αποτελούν καταπληκτική ευκαιρία Ευρώπη μα. Υπάρχουν πάρα πολλοί δημοσιογράφοι οι οποίοι περνάνε από φοβερές αντικσότητες, αντιμετωπίζουν πάρα πολλές δυσκολίες. Και ξέρετε ότι και η οικονομική κατάσταση αυτή τη στιγμή, η οικονομική συγκυρία πιέζει πάρα πολύ τον έντυπο τύπο. Υπάρχουν ε, πάρα πολλοί δημοσιογράφοι που εξαιτία τη οικονομική κατάσταση δεν μπορούν να είναι σε ελεύθεροι, θα μπορούσαν να είναι. Και γι' αυτό το λόγο με ανησυχεί πάρα πολύ το ζήτημα αυτό και είμαι σε συνεχή επαφή με τους εκδότες που έχουν να διαδραματίσουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για το ζήτημα αυτό και με τις οργανώσεις βέβαια που εκπροσωπούν και υπερασπίζουν τους δημοσιογράφους. Πολλοί βουλευτές επίσης αναφέρθηκαν στα δικαιώματα των παιδιών. Ήδη ανακοίνωσα ότι θα έχουμε σύντομα μία ανακοίνωση για τα δικαιώματα των παιδιών και στην ανακοίνωση αυτή θα προσπαθήσουμε να εξετάσουμε τα δικαιώματα των παιδιών σε σχέση με τη δικαιοσύνη. Αυτό θα αποτελέσει ένα από τα σημαντικά σημεία της ανακοίνωσης, γιατί πολύ συχνά τα παιδιά είναι το αδύναμο συμβαλόμενο μέρος, αν θέλετε, στις δικαστικές διαδικασίες και πολύ συχνά αποτελούν θύμα της δικαστικής διαδικασίας. Για να απαντήσω σε όλους αυτούς οι οποίοι αναφέρθηκαν στα παιδιά θα πω το εξή. Τα παιδιά δεν θα εμφανιστούν μόνο στην ανακοίνωσή μας για τα δικαιώματα των παιδιών, αλλά θα εμφανιστούν και στην ε, στρατηγική για τα άτομα με αναπηρία. Στρατηγική η οποία σύντομα θα εγκριθεί. Τα παιδιά με αναπηρία θα έχουν ε, μια ιδιαίτερη θέση στη γενικότερη αυτή στρατηγική για τα άτομα με αναπηρίες. Επίσης, έχουμε και όλο αυτό το γενικότερο ζήτημα της φτώχειας, της ένδυας. Η όλη συζήτηση πήγαινε ουσιαστικά για τους Ρωμά, πέρα από την πτυχή των, της διακρατικής μεταχείρισης, ήταν στην ουσία μια γενικότερη συζήτηση για την ε, φτώχεια, για την ένδυα. Και γι' αυτό το λόγο συνεργάζομαι με τον συνάδελφό μου επίτροπο Άντορο, είναι υπεύθυνο για το κοινωνικό ταμείο και με τον συνάδελφο Χάν, ο οποίος είναι υπεύθυνο για το περιφερειακό ταμείο. Θέλουμε ουσιαστικά να δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τους διαθέσιμους πόρους και υπάρχουν αρκετοί πόροι, αρκετά χρήματα, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ε, επενδύσει στην ε, καταπολέμηση της ε, φτώχεια και το λέω και το επαναλαμβάνω αυτό να γίνουν απαραίτητες επενδύσεις για την εκπαίδευση για τα παιδιά αυτά, γιατί δεν καταφέρουμε να επιλύσουμε το ζήτημα αυτό, δηλαδή το ζήτημα των παιδιών που δεν πηγαίνουν στα σχολεία, τα παιδιά τα οποία δεν καταφέρουν να έχουν πρόσβαση σε μια κατάρτιση. Σας λέω ότι σε 20 χρόνια θα συζητάμε τα ίδια πράγματα και θα πρέπει να επιλύσουμε τα ίδια προβλήματα. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε κατά αυτόν τον τρόπο. ετέθη ένα ζήτημα που είχε να κάνει με τη μεσολάβηση, αλλά πριν από αυτό θα ήθελα να αφαιρθώ στην παιδική πορνογραφία. Η συνάδελφος Μάλστρομ πρότεινε έναν κανονισμό για την προστασία των παιδιών online Το ζήτημα αυτό συζητάται από τους συνομοθέτες, από τα θεσμικά όργανα που συμμετέχουν στην νομοθετική διαδικασία και ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να βρεθούμε μια σωστή ισορροπία ανάμεσα στα δικαιώματα των παιδιών και την ελευθερία του διαδικτύου. Συχνά είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί αυτή η ισορροπία Πάντως εγώ πιστεύω ότι ε, κάθε φορά που αναφερόμαστε σε παιδιά και κάθε φορά που μιλάμε για εγκλήματα κατά των παιδιών, γιατί η παιδική πορνογραφία είναι έγκλημα κατά των παιδιών, ε, δεν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε διαφορετικά το φαινόμενο αυτό. Πολλές φορές στην περίπτωση αυτή, σε τέτοιες περιπτώσεις, αξίζει να μειωθεί εν μέρη και η ελευθερία του διαδικτύου. Α υποφέρει αν θέλετε λίγο η ελευθερία του διαδικτύου προκειμένου να καταφέρουμε να προασπίσουμε ένα τόσο σημαντικό ε, θεμελιώδες δικαίωμα όπως ε, τα δικαιώματα των παιδιών. Και πιστεύω ότι απαντώ κατά αυτόν τον τρόπο και στην ερώτηση της κυρίας Βάλεαν. Το ζήτημα της ελευθερίας του διαδικτύου είναι κάτι το οποίο απασχολεί όλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ξέρετε ότι και εγώ είμαι στη δική σας αστικά την πλευρά, χρειαζόμαστε να έχουμε την ελευθερία αυτή, θα πρέπει όμως να καταφέρουμε να θεσμοθετήσουμε και την ε, περίπτωση εκείνη όπου η ελευθερία διαδικτύου μπορεί να βαίνει κατά των δικαιωμάτων των παιδιών. Ξέρετε επίση ότι η συνάδελφος, ε, η συνάδελφος Κρούς ασχολείται με το ζήτημα της ουδετερότητας ε, και της διαμεσολάβησης στο οποίο αναφερθήκατε. Θα βρεθεί λύση σε κοινοτικό επίπεδο. Επίσης, την προηγούμενη εβδομάδα ένας Αμερικανός συνάδελφος έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Μου είπε ότι εσείς οι Ευρωπαίοι έχετε δίκιο Κάθε φορά που προσπαθείτε με το δικό σας τρόπο να διευθετήσετε το ζήτημα της ουδετερότητας, το ζήτημα του net neutrality. Όσον αφορά τις Βρυξέλλες 2α και την Jugendamt. Επανερχόμαστε εδώ πέρα σε ένα ζήτημα το οποίο έχουν ε, αναφέρει πάρα πολύ στο παρελθόν. Ποια είναι τα όρια της επικορικότητας και πού ξεκινά η ε, ευρωπαϊκή ευθύνη. Ως Επίτροπος, αυτό μπορώ να κάνω, είναι αυτό που με επιτρέπουν ουσιαστικά οι συνθήκες να κάνω. Οι συνθήκες είναι αυτές που δίδουν την απάντηση. Την προηγούμενη εβδομάδα δημοσιεύθηκε ένα Μέκουμ, ένας οδηγός για την εφαρμογή του χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η εφαρμογή του χάρτη αυτού συνδέεται με τις συνθήκες ουσιαστικά εφαρμόζεται όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο επεξεργάζονται κοινοτική νομοθεσία. Επομένως, σε όλη αυτή τη νομοθετική διαδικασία εφαρμόζεται ο χάρτης των θεμελιωδών και εφαρμόζεται επίσης και όταν οι ευρωπαϊκοί αυτοί κανόνες μεταφέρονται στην εθνική πρακτική, στην εθνική νομοθεσία. Διαβάστε σας παρακαλώ πολύ τι έγραψα σε αυτό το βαντεμέκιου, γιατί πραγματικά εκεί πέρα εξηγώ πολύ καλά πού μπορούμε να λάβουμε δράση και πού όχι. Θα ήταν παραπλανητικό πιστεύω το να πούμε στους πολίτες ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί πλέον να αναλάβει δράση παντού. Όχι, εξακολουθεί να ισχύει η αρχή της επικουρικότητας. Επανέρχομαι τώρα στη Jugendamt. Δεν θα πω ότι δεν μπορώ να δώσω καμία απάντηση στο ζήτημα αυτό. Είδα την απάντηση που δώσαν οι γερμανικές αρχές για το ζήτημα. Και αναφέρονται εδώ πέρα στα συμφέροντα, τα καλύτερα δυνατά συμφέροντα του παιδιού. Από όσο θυμάμαι λοιπόν, θα πω κάποια πράγματα, Ένα 13% των γάμων σήμερα είναι μεικτή γάμη. Δηλαδή οι γονείς είναι διαφορετική εθνικότητας και πολύ συχνά ζουν και σε άλλη χώρα, σε άλλο κράτος μέλος. Πιστεύω ότι κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να έχει και τους δυο του τους γονείς. Και αν έχουμε ένα μεικτό γάμο, τότε το παιδί αυτό έχει δικαίωμα και στους δύο πολιτισμούς ή και σε ένα τρίτο πολιτισμό αν ζουν σε μια άλλη χώρα διαφορετική από αυτή των, της των, γονέων. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Δεν μπορούμε στα πλαίσια του περιβάλλοντος ελεύθερης μετακίνησης και της ελεύθερης κυκλοφορίας να σκεφτόμαστε διαφορετικά, γιατί το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας αποτελεί δικαίωμα κάθε πολίτη. Επομένως, θα πρέπει να είναι και ένα δικαίωμα του παιδιού, θα πρέπει το παιδί μάλλον να έχει δικαίωμα σε περισσότερους πολιτισμούς και περισσότερες γλώσσες. Επίσης, πολύ σωστά οι αρχές προσπαθούν να ισορροπήσουν κάπως τα πράγματα. Ενδεχομένω ένας από τους δύο γονείς να υπερβάλλει κάπως τη στάση του και τη συμπεριφορά του. Οι αρχές προσπαθούν να δουν κάθε φορά ποια είναι τα δικαιώματα του παιδιού και το δικαίωμα του παιδιού όμως δεν μπορεί να είναι το παιδί το οποίο ζει στη Γερμανία να έχει απλώς πρόσβαση στη γερμανική γλώσσα και έγραψα μάλιστα και μια επιστολή απευθυνόμενη στις γερμανικές αρχές και του ζήτησε να μου δώσουν περισσότερες πληροφορίες για την υπόθεση αυτή. Yeah. Uh, why don't... Τώρα, για ποιο λόγο οι πολίτες δεν λαμβάνουν απαντήσεις πιο γρήγορα. Γιατί μα και οι ευρωβουλευτέ δεν λαμβάνουν απαντήσει ε, νωρίτερα και εσεί ίδιοι παραπονιέστε. Συχνά η απάντηση προς ένα πολίτη δεν δίνεται από έναν μόνο επίτροπο. Με έχει απασχολήσει το ζήτημα αυτό γιατί έλαβα πολλά παράπονα και συχνά αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι μου φτάνει ένα παράπονο, μια καταγγελία, ένα ερώτημα, αλλά πρέπει να διευκρινίσω κάπως τα πράγματα προκειμένου να δοθεί μια απάντηση από τι υπηρεσίε μου οι οποίε θα πρέπει να συνεργαστούν με τρει-τέσσερι άλλου επιτρόπους που ε, έχουν και αυτοί μια σχετική αρμοδιότητα για το ζήτημα και πρέπει να συνεργαστούν και αυτοί με τη σειρά του με την νομική υπηρεσία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα πράγματα είναι πιο πολύπλοκα. Τελικά τα πράγματα είναι πιο πολύπλοκα από ό,τι φαίνεται. και γι' αυτό το λόγο πολλές φορές απαιτείται πολύ περισσότερος χρόνος από ότι θα ήταν αποδεκτό από τους πολίτες προκειμένου τους δοθεί μια απάντηση και αυτό σαφώς είναι ένα πρόβλημα γιατί ε, δεν τον ενδιαφέρει τον πολίτη το γεγονός ότι πρέπει τέσσερις επίτροποι να ενσκύψουν στο πρόβλημά του και ολόκληρη η υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο πολίτης αυτό το οποίο θέλει είναι μια απάντηση. Και γι' αυτό το λόγο τροποποίησα το σύστημα βάσει του οποίου μπορεί ο πολίτης να απευθυνθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σα είπα ότι έχει δημιουργηθεί μια νέα θηρίδα, το Europe Direct Network, μέσω, του οποίου, μέσω, μέσω της οποίας ο πολίτης μπορεί να απευθύνεται άμεσα και γρήγορα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μία θηρίδα θα πρέπει να είναι αυτή στην οποία να απευθύνεται ο Ευρωπαίος πολίτης και δεν θα πρέπει να νοιάζει το πολίτη στη συνέχεια για τον το δρόμο που θα ακολουθήσει το αίτημά του. Προσπαθώ να μεταρρυθμίσω λοιπόν όλο αυτό το σύστημα. Σίγουρα το εγχείρημα δεν είναι εύκολο και σίγουρα τα πράγματα δεν μπορούν να κινηθούν πάρα πολύ γρήγορα. Νομίζω ότι απάντησα πάνω κάτω σε όλες τις ερωτήσεις που έθεσαν οι Ευρωβουλευτές. Ευχαριστώ. Το αξίζατε με το παραπάνω το χειροκρότημα. Ευχαριστούμε την κυρία Ρέντινγκ για την ε, συνεισφορά της. Ελπίζουμε το επόμενο ραντεβού που, προδι... που μας εξαγγείλατε πάνω κάτω και ελπίζω ότι θα τα ξαναπούμε σύντομα και θα τύχει η Επιτροπή μας μεγαλύτερης προσοχής. Ένα διαδικαστικό για την ημερήσια διάταξη τώρα. Εμείς αύριο θα συνεχίσουμε στα από τα σημεία που διακόψαμε σήμερα την αναφορά δηλαδή που ακούσαμε με την τοποθέτηση της κυρίας που είναι υπογράφουσα. Αύριο από τις, 10 θα συνεχίσουμε.